Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ να φορέσετε τα κουστικά σας, να μην καπνίζετε στην αίθουσα. Αξιότιμοι καλεσμένοι, είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ σήμερα να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ. Ονομάζομαι Μίρτσια Διακόνου, είμαι από την ε, ε, Ρουμανία και θα αναλάβω την Προεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα ε, μπορούμε να κηρύξουμε την έναρξη της συνεδρίασης της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά και χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω τόσα πολλά μέλη των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων εξ ονόματος ε, εμού και των άλλων μελών της Επιτροπής Πολιτισμού που δεν μπορούσαν σήμερα να είναι εδώ μαζί μας. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Η εκδήλωση αυτή οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να μπορέσουμε να τιμήσουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018. Ο στόχος της ε, ε, σημερινής συνεδρίασης είναι να συζητήσουμε διάφορα θέματα που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς να μιλήσουμε για τον ε, αντίκτυπο που θα έχει το ευρωπαϊκό αυτό πολιτιστικό έτος και βεβαίως να δούμε και πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για καλές πρακτικές που έχετε συλλέξει εσείς σε εθνικό επίπεδο. Και βεβαίως να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για την πολιτιστική κληρονομιά και στο μέλλον. Στα πλαίσια της τελευταίας συνάντησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής είχαμε αποφασίσει ότι θα έχουμε δύο τμήματα στην σημερινή συνάντηση ε, και ταυτόχρονα γίνονται τρεις διαφορετικές συνεδριάσεις σε τρία πάνελ. Ένα που ασχολείται με τον πολιτισμό και την ταυτότητα, ένα με την διατήρηση, συντήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ένα τρίτο που ασχολείται με την ε, πολιτιστική κληρονομιά και την εκπαίδευση. Αύριο θα γίνει μια κοινή ολομέλεια με όλους τους ε, συμμετέχοντες έτσι ώστε να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της σημερινής ημέρας. Το πάνελ λοιπόν είναι ανοιχτό, οπότε μπορείτε όλοι να πάρετε το λόγο και να μιλήσετε. Αύριο θα ακούσουμε μόνο τους εθνικούς βουλευτές, κάποιους ευρωβουλευτές και κάποιους επιλεγμένους ομιλητές. Γι' αυτό σήμερα καλό είναι να πάρετε το λόγο εφόσον το θέλετε Έχουμε βουλευτές από, τις, ε, ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια σήμερα μαζί μας, έχουμε συναδέλφου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε ειδικού, εμπειρογνώμονε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την UNESCO, εθνικούς συντονιστέ ε, του Ευρωπαϊκού Έτου, τη Πολιτιστική Κληρονομιά και εκπροσώπους της Κοινωνία των πολιτών και οργανώσεων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, χαίρομαι που ε, δεχτήκατε όλοι να είσαστε παρόντες σήμερα στην συνάντηση αυτή. Κάποιοι εμπειρογνώμονε μα είπαν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή οδηγία για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, γιατί έτσι θα ήταν τα πράγματα πολύ πιο απλά. Βεβαίω αυτό αλήθεια είναι, αλλά δυστυχώ είναι αδύνατο. Το ξέρετε, γιατί ο πολιτισμός, η πολιτιστική, η πολιτιστική κληρονομιά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν μπορεί να τη ρυθμίσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα θέματα τους ή άλλως είναι ιδιαίτερο ευαίσθητα και συνδέονται πάρα πολύ με την εθνική ταυτότητα των κρατών. Πριν λοιπόν συζητήσουμε το οτιδήποτε, πρέπει να θεωρήσουμε ότι το θέμα αυτό θα μπορέσει να παραμείνει σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Βεβαίω, το Ευρωπαϊκό Έτο πολιτιστική Κληρονομιάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί πολλοί εμπειρογνώμονε, πολλοί ειδικοί ε, συνέρχονται για να συζητήσουν όλα αυτά τα σημαντικά θέματα που απτώνται τη πολιτιστική κληρονομιάς. Όλα αυτά τα θέματα περιλαμβάνονται σε 10 συγκεκριμένε πρωτοβουλίε τι οποίε θα ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ήμουνα εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι διάφορε αυτέ πρωτοβουλίε και μάλιστα εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερω για το πόσο ει βάθους μελέτησαν οι συμμετέχοντε στα θέματα αυτά. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο συστάσει μπορεί να, να προτείνει για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κληρονομιά. Για να γίνουν αυτέ αυτές οι συστάσει αποτελέσματα απτά χρειαζόμαστε εσά, του εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων οι οποίοι θα προωθήσετε τα μηνύματα αυτά στις χώρες σας. Εγώ ε, ζήτησα από την ε, νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου να είναι μαζί μας. Ο Τζοβάνι Μεντόλα είναι μαζί μας σήμερα από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για να μπορέσει να μας συμβουλεύσει για την ευρωπαϊκή κληρονομιά από την νομική πλευρά. Οπότε προτείνω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα θα μας κάνει μια παρουσίαση για τη δομή του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς και θα μας παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα συζητήσουμε σήμερα μαζί σας. Την ε, παρουσίαση θα μας την κάνει η κυρία Ερμήνια Σκιακιτάνο και βεβαίως ε, οι υπόλοιποι συνάδελφοι από τις άλλες γενικές διευθύνσεις θα πάρουν το λόγο αργότερα. Μετά θα κάνουμε άλλη μια συζήτηση για άλλα θέματα που ασχολούνται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα μιλήσουμε κυρίως για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη να υπάρξει βιώσιμος τουρισμός. Ε, προτείνω λοιπόν μετά από τις παρουσιάσεις που θα ακούσουμε να κάνουμε μία ε, συζήτηση έρωτα-απαντήσεων, να ακούσουμε παραδείγματα ε, καλών πρακτικών και στο τέλος θα εξαχθούν κάποια συμπεράσματα, τα οποία όμως αύριο θα παρουσιαστούν στην Ολομέλεια. Πριν δώσουμε τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα οργανωτικά. Καταρχάς, το αργότερο στις 6 και 20 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει γιατί πρέπει να πάμε στο κοκτέιλ. Έχουμε ε, σήμερα ε, διερμηνία στις 23 γλώσσες τη Ένωση και η συζήτηση μεταδίδεται ζωντανά και στο διαδίκτυο. Οπότε περνάμε αμέσως στην κυρία Σκιακιτάνο, η οποία θα μας παρουσιάσει το γενικό πλαίσιο και τις 10 πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Uh, thank you, me the floor. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας και να σας ε, παρουσιάσω αυτή την εξαιρετική εμπειρία που ήταν η, διοργάνωση και η διαχείριση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. Να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για το μόνο ευρωπαϊκό έτος κατά τη διάρκεια της αιτίας της Επιτροπής Juncker. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστή για την πολιτική της κληρονομιά. Θα σας πω, ε, θα σας μιλήσω για τον τεράστιο αριθμό ε, σημείων πολιτικής κληρονομιάς που έχουμε στην Ευρώπη. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη με πολιτικά κέντρα, πολιτικούς εμπειρογνώμονες κλπ. Όμως ε, η πολιτική κληρονομιά δεν είναι κάτι το παθητικό. Πρέπει συνεχώς ε, να είναι κανείς δραστήριος για να μπορέσει να τη μεταλαμπαδεύσει στις επόμενες γενιές. Δεν μπορούμε να τη θεωρούμε δεδομένη την πολιτική κληρονομιά. Η πολιτική μας κληρονομιά ιδιαίτερα σήμερα περιλαμβάνει αρχές, διδάγματα και μνήμες πάρα πολύ σημαντικές για την σημερινή Ευρώπη αλλά και για την οικοδόμηση της μελλοντικής Ευρώπης. Γιατί η πολιτική κληρονομιά περιλαμβάνει την ιστορία και τα διδάγματα που έχουμε λάβει από τις επιτυχίες μας, αλλά και από τις αποτυχίες μας. Για παράδειγμα, από τις συγκρούσεις ή από τους πολέμους που λάμβαναν χώρα στην Ευρώπη παλιότερα. Πολύ σημαντικά μαθήματα και γι' αυτό το λόγο Στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτικής Χρονιάς, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είχαν θέσει ως ε, στόχο να τονιστεί η σημασία της πολιτικής κληρονομιάς ως ε, στοιχείο συνειδητοποίησης της ε, κοινή μας ιστορίας και των κοινών μας αρχών και ως ένα σημαντικό στοιχείο κοινή ταυτότητας. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε ε, την αντιμετώπιση της ε, πολιτικής χρονομιάς ως ε, κοινού πλούτου. Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς μπορούμε να την προστατέψουμε καλύτερα και να μπορέσουμε να την περάσουμε στις επόμενες γενιές, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στη σημερινή κατάσταση η διαχείριση Τη πολιτική χρονομιά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, παγκοσμιοποίηση, ψηφιοποίηση, πολλέ προκλήσει. Το πρόβλημα επίση μετάδοση τη γνώση από τη μία γενιά στην επόμενη κλπ. Γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε να αναλάβουμε δράσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να στηριχθεί ο τομέα και να αντιμετωπιστούν αυτέ τι προκλήσει. Ε, άλλωστε, ε, ε, κληθήκαμε και από τους ε, ε, ίδιους τους ε, πολίτες να αναλάβουμε, ε, αναλάβουμε δράση. το Ευρωβαρόμετρο στο τέλος του 2017 αναφέρει πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχήν το ότι για τους Ευρωπαίους η πολιτική κληρονομιά είναι σημαντική. Το 80% όσων ερωτήθησαν είπαν ότι είναι σημαντική η πολιτική κληρονομιά τους και για τις κοινότητε του. Το 80% επίσης ε, είπαν ότι είναι σημαντική η πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 82% είναι πεπισμένοι ότι η πολιτική κληρονομιά είναι σημαντική γιατί δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. 82% θεωρούν τους αυτούς τους περήφανους για την πολιτική τους Και επίσης το 70% είναι περήφανοι για την πολιτιστική κληρονομιά που δεν ανήκει στην επικράτεια της χώρας τους. Δηλαδή, πολιτιστική κληρονομιά που εντοπίζεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν ε, δείτε ότι αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως ε, ε στοιχείο ένδειξη ε, του ανήκειν στην κοινή Ευρώπη. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η πολιτική μας κληρονομιά είναι ένα σημείο στο οποίο συνδέεται το παρελθόν με το μέλλον. Δεν πρόκειται για κάτι που έχει απαρχαιωθεί και ανήκει στο παρελθόν, αλλά είναι σημαντική πηγή και για το μέλλον μας. Ε, δημιουργήσαμε λοιπόν μια εκστρατεία και εργαλεία, ένα site στο ίντερνετ, μια, μια ηλεκτρονική εφημερίδα, ένα newsletter. Και σήμερα εδώ ιδιαίτερα σε αυτό το πάνελ θα εξετάσουμε κάποιες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στο πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον τομέα αυτό ε, της προστασίας της πολιτικής μας κληρονομιάς. Μερικά νούμερα για το τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Μέσω διαφόρων, ε, ε της οργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Ε, και με άλλα μέσα. Ε, ένας πολύ μεγάλος αριθμό εκδηλώσεων οργανώθηκαν, πάνω από 11.000 σε όλη την Ευρώπη. Ε, η εκδήλωση λήξης του έτους θα λάβει χώρα στη Βιέννη σε 6 και 7 Δεκεμβρίου και με εκείνη την ευκαιρία θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και θα αναφέρουμε και τα οριστικά τελικά νούμερα. 6,2 εκατομμύρια άτομα ήταν το κοινό μας μέχρι σήμερα με ένα μεγάλο αριθμό project σχεδίων που χρηματοδοτούνται και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο μέσω της, του χαρακτηρισμού ότι ανήκουν στο έτος αυτό. Πάνω από 900 τέτοια project στην Ευρώπη και πάνω από 7.900 project σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, 229 project που ε, χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη με ένα ειδικό προπολογισμό ο οποίος συμπεριελήφθη στη νομική βάση αυτού του ε, έτους Ευρωπαϊκής Κοινωνίας. Αυτά τα 29 σχέδια είχαν ε, δώσει έμφαση στην αίσθηση του ανήκειν στην ευρωπαϊκή διάσταση πολιτικής κληρονομιάς και στην δυνατότητα μέσω της πολιτικής κληρονομιάς να τονιστεί η σημασία του να ανήκει κανείς στην Ευρώπη. Όμως, είχαμε και άλλου τύπου χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. Για παράδειγμα, από το πρόγραμμα Horizon 2020-2020, έχω κάποια νούμερα, αλλά οι συνάδελφοί μας θα σας πούνε περισσότερα πράγματα. και άλλου τύπου χρηματοδότηση μέσω του Erasmus Plus, το Ευρώπη για τους πολίτες, τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία συνοχής κλπ. Συλλογική εργασία λοιπόν. Όμως το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτικής Χρονομιάς δεν είναι το άθροισμα κάποιων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια Το σημαντικό κατά τη διάρκεια αυτού του έτους είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε, προστατεύουμε ε, και συντηρούμε την πολιτική μας κληρονομιά. Να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό το λόγο, στο έτος πολιτικής κληρονομιάς δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο τι θα αφήσουμε στο μέλλον, ε, τι κληρονομιά θα αφήσουμε στο μέλλον. Και όπως με ένα παγόβουνο, αυτή η κληρονομιά είναι ενδεχομένως λιγότερο ορατή είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας όπως η μεγαλύτερη μάζα του παγόβουνου αλλά πάρα πολύ σημαντική. Και ποια είναι λοιπόν τα θεμέλια αυτής της κληρονομιάς που θα αφήσει το έτος πολιτικής κληρονομιάς. Τα θεμέλια αυτά ε, σχετίζονται άμεσα με την σοβαρότατη συζήτηση που ε, ξεκίνησε το 2014 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία συμμετείχαν όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο, η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και αντιπρόσωποι των κρατών μελών των εθνικών διοικήσεων. Αυτή η συζήτηση διαμόρφωσε ένα τελείως καινούριο τρόπο να βλέπουμε την πολιτική μας κληρονομιά. Για παράδειγμα, όλοι πλέον έχουμε συμφωνήσει ότι η πολιτική κληρονομιά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ολιστικά, ολιστικά ε, εξετάζοντας όλες τις πτυχές ε, ε, άειλη και ψηφιακή. Εγώ για παράδειγμα προέρχομαι από το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτικής Ονομιάς και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό που καταφέραμε να φέρουμε μαζί ε, όλες αυτές τις προσεγγίσεις σε ε, μία ενιαία αντιμετώπιση. Μία άλλη επιτυχία που προέκυψε από αυτή την συζήτηση ήταν το εξής. Η πολιτιστική κληρονομιά ε, είναι ένας πόρος, ένας, μια πηγή πλούτου οφέλει ωφελεί το περιβάλλον, ωφελεί την οικονομία, ωφελεί την κοινωνία στο σύνολό τη και σίγουρα την πολιστική ποικιλομορφία. Όμως, για να φτάσουν όλα αυτά τα ωφέλη στους δικαιούχους τους, ε, δεν μπορούμε απλώς να δρούμε παθητικά. Πρέπει να ε, παίρνουμε πρωτοβουλίες και μάλιστα με έναν τρόπο σφαιρικό, εξετάζοντας όλες τις διαφορετικές πολιτικές τις οποίες η πολιτική κληρονομιά είναι σημαντική συνιστόσα. Για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πολιτική κληρονομιά είναι συστατικό διαφόρων πολιτικών της περιβαλλοντικής πολιτικής, της πολιτικής έρευνας, του τουρισμού βέβαια και βέβαια σημαντική συνιστόσα και της παιδείας, εκπαίδευσης. Επίσης, τα διαστατικά ταμεία χρηματοδοτούν ε, πολλές πτυχές της πολιτικής κληρονομιάς ως ε, εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης ε, και συνοχής. Αν όλα αυτά δεν κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, ε, θα κατακαιρματιστούμε και θα πάψουμε να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον. Μια μελέτη η οποία χρηματοδοτήθηκε από, ένα από το πρόγραμμα Culture πρόκειται για τη μελέτη «Η πολιτική κληρονομιά είναι σημαντική για την Ευρώπη». Παρακαλώ πολύ διαβάστε την. Το consortium μου, το οποίο ήταν η Europa Nostra ανέλησε ε, πάνω από 200 ε, μελέτες για την πολιτική κληρονομιά και υπογραμμίζει τη σημασία ε, να αντιμετωπίσουμε την πολιτική κληρονομιά με έναν τρόπο πιο δραστήριο και ολιστικό σφαιρικό. Πώς αυτό θα γίνει πράξη στην, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γίνεται πράξη μέσω της αρχής του mainstreaming, της ένταξη δηλαδή της πολιτική χρονομία, οριζόντια σε όλες τις ε, συναφείς πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό άλλωστε τονίστηκε και στην νομική βάση του Ευρωπαϊκού της Πολιτικής Κληρονομιάς, όπου ζητείται από την Κομισιόν να εργαστεί καλύτερα, πιο οριζόντια και να εξερευνήσει όλες τις δυνατές συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών. Καταλαβαίνετε πόσο περίπλοκο είναι κάτι τέτοιο. Για να δώσει αποτελέσματα αυτή η προσπάθεια, δημιουργήσαμε ένα πολύ περίπλοκο μοντέλο διακυβέρνησης. Αυτή η δομή αναφερόταν ήδη στην νομική βάση του Ευρωπαϊκού Έτος Πολιτικής, ανα... Ε, ε, το Ευρωπαϊκό Έτος το διαχειρίζεται σε επίπεδο κρατών μελών μια ομάδα εθνικών συντονιστών που ορίζονται από τα κράτη-μέλη. Αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτική κληρονομιά εμπίπτει στην αρχή τη επικουρικότητα, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά δίνεται η δυνατότητα να συντονίσουμε τι δραστηριότητε σε ευρωπαϊκό πεδίο και ιδιαίτερω να προβούμε σε ανταλλαγέ καλών πρακτικών, υβέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών συντονιστών. Επίση, έχουμε εννέα συνδεδεμένε χώρε, δεν περιοριστήκαμε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχουν και άλλες εννέα χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης ε, συμμετέχει πλήρως, συμμετέχει και στην Επιτροπή των Εθνικών Συντονιστών. Επίσης είναι παρόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κ. Διάκονο συγκεκριμένα σε μια άλλη πολύ σημαντική επιτροπή που δημιουργήθηκε που είναι η επιτροπή στην οποία έχουν φωνή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του τομέα της πολιτικής κληρονομιάς. Είναι οι βασικές πλατφόρμες, οι βασικοί φορείς, τα βασικά δίκτυα που ασχολούνται με θέματα πολιτικής κληρονομιάς. Και βέβαια διεθνεί οργανώσει όπω η Βουλή τη Ευρώπη, η UNESCO, ε, η ΕΚΡΟΜ κλπ. Βέβαια, ε, δικτύα όπως το ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις κλπ. είναι επίσης μέλη αυτής της Επιτροπής των εμπλεκομένων φορέων, των stakeholders. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης εμπλέκονται. Η Γενική Διεύθυνση ε, Πολιτισμού και Παιδείας, επίσης εγώ την εκπροσωπώ για παράδειγμα, Λαμβάνουμε υπόψη επίσης ε, το σημαντική, τη σημαντική πτυχή του αθλητισμού και της νεολαίας και αυτό αποτελεί τμήμα της γενικής μας διεύθυνσης. Όπως βλέπετε όμως έχουμε και άλλες γενικές διευθύνσεις οι οποίες συνεργάζονται μαζί μας. 19 συνολικά υπηρεσίες συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτικής Ανάπτυξης. Το input των ε, εμπλεκομένων φορέων μέχρι τώρα είναι ότι ε, το ευρωπαϊκό έτος ε, θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα συμμετέχουν με πολύ ενθουσιασμό. Για να κινηθούμε προς ένα κοινό στόχο, προς ένα κοινό σχέδιο μέχρι το τέλος του χρόνου, τι κάναμε, εντοπίσαμε τις, αυτό που αποκαλούμε 10 ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες για όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. θα σχολιάσουμε τις ε, πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με το αντικείμενο αυτού του πάνελ. Όμως ε, θα δείτε δίπλα στους ε, τίτλους των πρωτοβουλειών τα αρχικά των γενικών διευθύνσεων που εμπλέκονται. Ευρωπαϊκό ιδιόλεκτο όλα αυτά. Οι δέκα αυτέ τι ευρωπαϊκέ πρωτοβουλίε ε, διαρθρώνονται σε τέσσερι πυλώνε. Πυλώνα τη ε, προσήλωση, τη βιωσιμότητα, τη προστασία και τη καινοτομία. Στον πρώτο πυλώνα εστιάζουμε τις προσπάθειές μας ιδιαίτερα στην καινούργια γενιά που είναι και η διάδοχή μας, η διάδοχη των παλιότερων γενιών, η κληρονόμη μας. Εδώ έχουμε την εκπαίδευση, την διδημοποίηση, τα σώματα αλληλεγγύης, ε, τους εθελοντές και όλα αυτά. Συνεργασία λοιπόν σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο νέων. Ο πυλώνας της βιωσιμότητας, ο δεύτερος πυλώνας, εξετάζει πιο πολύ αυτά που έλεγα πριν, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η παρέμβαση της πολιτικής κληρονομιάς δημιουργεί, μια, ε, δημιουργεί βιώσιμες ε, συνέπειες. Εδώ συνεργαζόμαστε με τη Διεύθυνση Grow, τη Γενική Διεύθυνση του ε, Περιβάλλοντος. Η, ο συνάδελφος σας πει πολλά για αυτά το πράγμα, με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας, επίσης θα ακούσετε ένα εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας αργότερα και έχουμε βέβαια και τους άλλους δύο πυλώνες προστασίας και καινοτομίας. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτούς. Καταρχήν όμως να ξεκινήσω από τον πυλώνα της βιωσιμότητας. Θέλω να σας παρουσιάσω μία από τις πιο βασικές μας δράσεις που είναι ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός. Όπως ε, σας είπα, ο τουρισμός είναι ένα σημαντικός μοχλός τοπικής ανάπτυξης, αλλά γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός θα πρέπει να τη χάνει διαχείριση ε, με βιώσιμο τρόπο. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να βλάψει την πολιτική κληρονομιά. Και γι' αυτό το λόγο δώσαμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μια σειρά κρατών μελών που έχουν δημιουργήσει μια ομάδα που συζητά το θέμα και εκδίδει συστάσεις για το βιώσιμο πολιτιστικό ε, τουρισμό, συστάσεις που θα είναι ολοκληρωμένες και έτοιμες στο τέλος του χρόνου. Θα, ένα προσχέδιο αυτών θα παρουσιαστεί στη Βιέννη 6 και 7 Δεκεμβρίου. Στις 25 και 26 Οκτωβρίου έγινε μια παρουσίαση στην ΠΑΦΟ με κάποια πρώτα στοιχεία για τα πορίσματα αυτής της Επιτροπής. Μετά, ο άλλος πυλώνας της προστασίας. Ε, εδώ θέλω να προσέξουμε μία πρωτοβουλία που είναι η χρήση, η σωστή χρήση της πολιτικής κληρονομιάς αναπτύσσοντας προδιαφές ποιότητας για την παρέμβαση στην πολιτική κληρονομιά. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι μια περιοχή αριστείας σε ό,τι αφορά την προστασία της πολιτικής κληρονομιά. Όμως για πολύ καιρό δεν έχουμε συμφωνήσει ε, επί βασικών αρχών και μάλιστα δυναμικών αρχών που θα αλλάζουν με το χρόνο. Γι' αυτό το λόγο είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί για το τι σημαίνει ποιότητα τι σημαίνει ανάπτυξη ποιοτικών προδιαγραφών, τι σημαίνει αυθεντικότητα για την Ευρώπη σήμερα όταν παρεμβαίνουν στην πολιτική κληρονομιά. Και επίσης πόσο σημαντική είναι αυτή η αυθεντικότητα, πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε για προγραφές ποιότητας δεδομένου ότι στην πολιτική κληρονομιά χρησιμοποιούνται και ευρωπαϊκοί πόροι. Ιδιαίτερα αν θέλουμε να εντάξουμε την πολιτική κληρονομιά σε διάφορες πολιτικές έτσι ώστε να χρησιμοποιεί ποσά από διάφορα ταμεία και εργαλεία τα οποία όμως μπορεί να έχουν διαφορετικό αρχικό στόχο τότε υπάρχει ο κίνδυνος ε, να δοθεί λιγότερη σημασία στις αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν την πολιτική κληρονομιά. Γι' αυτό το λόγο, και γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια εισήγηση του κ. Διάκονου το 2015 είχε υπογραμμίσει την σημασία να συζητήσουμε τι σημαίνει ποιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, ζητήθηκε από την Κομισιόν στην ε, νέα γενιά των ε, διαστατικών ταμείων να συμπεριλάβει ένα ε, πρόγραμμα ποιότητας και προδιαφών ποιότητας οριζόντια. Αυτό αποτελεί τμήμα πρωτοβουλία τη ε, διάσκεψη που διοργάνωσε η Λετωνική Προεδρία του 2015. Εκεί συζητήθηκε το θέμα της καλύτερης συνεργασίας, συνέργειας ανάμεσα στην διατήρηση της πολιτικής οικονομιάς και την σύγχρονη, στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό ε, σχεδιασμό. Το Ευρωπαϊκό Έτο Πολιτική Χρονομιά, λοιπόν συμπεριέλαβε μεταξύ των στόχων του την πρόθεση της συζήτηση, ανταλλαγή, ε, και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την ποιοτική συντήρηση και διατήρηση της πολιτική χρονομιά και του ιστορικού περιβάλλοντος. Το Συμβούλιο υπογράμμισε πρόσφατα τη σημασία όλων αυτών στα συμπεράσματά του υπογράμμισε την ε, σημασία της ένταξης της πολιτικής ονομιάς σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ότι θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ποιες, ποιες είναι οι αρχές που διαπούν την πολιτική κληρονομιά. Κάλεσε την Κομισιόν συγκεκριμένα το Συμβούλιο όταν εφαρμόζει και ε, αξιολογεί τις διάφορες ε, προτάσεις να λαμβάνει υπόψη το πώς τα σχέδια αυτά επεμβαίνουν ε, στην βελτίωση, διατήρηση και την προστασία της ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας και ιδιαίτερα στην ανάγκη για ποιοτικέ ε, κατευθυντήρες γραμμές για να εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, βλάπτουν την πολιτική κληρονομιά και τις αρχές της. Γι' αυτό το λόγο, στο πλαίσιο του ΙΚΟΜΟΣ, ε, μάλλον με συντονιστικό όργανο το ΙΚΟΜΟΣ δημιουργήσαμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Όπω καταλαβαίνετε ότι αυτά, αυτά τα θέματα μπορούν να συζητηθούν μόνο μεταξύ ειδικών. Στόχος της ομάδας είναι τα αποτελέσματα να είναι ε, προσβάσιμα και κατανοητά ακόμα και από μη ειδικούς. Ακριβώς διότι προωθούμε μια συμμετοχική διαχείριση της πολιτικής κληρονομιάς. Εδώ πέρα έχουμε το χρονοδιάγραμμα. Έλαβαν χώρα διάφορες συναντήσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων. Έχουμε ένα πρώτο προσχέδιο εγγράφου, το οποίο θα συζητηθεί στις 22 και 23 Νοεμβρίου στη Βενετία. Σύντομα δηλαδή. Μετά από αυτή τη συζήτηση πρόθεση της Κομισιόν είναι να ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση για το θέμα αυτό. Επίσης είναι σημαντικό και αυτό δείχνει την, τον εσωτερικό συντονισμό μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Το, ορίζο, το πρόγραμμα Horizon 2020 το 2009 θα στηρίξει τη δημιουργία ε, μιας κοινωνικής πλατφόρμας εμπειρογνωμόνων και εμπλεκομένων φορέων που θα συνεχίσουν τι συζητήσει για αυτό το θέμα. Αφού έχουμε λοιπόν το πρώτο βασικό έγγραφο για τις ε, αρχές ε, ποιότητας, ε, το θέμα θα συνεχίσει να συζητείται στο πλαίσιο του Ορίζον 2020. This is the, these are the dates of the conference and Έχουμε λοιπόν εδώ τις ημερομηνίες των συναντήσεων και κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τους διαγωνισμούς προκειμένου να συσταθεί αυτή η κοινωνική πλατφόρμα 14 δηλαδή Μαρτίου του 19. Άλλη μια σημαντική πρωτοβουλία είναι η πρωτοβουλία Heritage at Risk προκειμένου να προστατεύσουμε ε, μνημεία συγκεκριμένα πολιτιστικής ε, κληρονομιάς εντός της πρωτοβουλίας αυτής όπως βλέπετε και στον τίτλο κοιτούμε υπό δύο οπτικές. Καταρχάς, την ε, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την διαχείριση του κινδύνου ή στα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για την καταπολέμηση Υπάρχει ήδη ένα νομικό πλαίσιο, αλλά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που είναι ιδιαίτερα τα πρώτα τρία έγγραφα που έχω τοποθετήσει εδώ αποσκοπεί στην αποφυγή της εξαγωγής της παράνομης εξαγωγής προϊόντων και στοιχείων της ε, πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εξαγωγής δηλαδή εκτός του εδάφους Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράνομης εμπορίας. Οι διάφορες καταστροφές που έχουν βεβαίως συμβεί στην Μέση Ανατολή μας οδηγούν και σε μια ανάγκη προστασίας διαφορετικής πολιτιστικής κληρονομιάς από άλλα μέρη του κόσμου που επίσης διακινούνται παρανόμως. Εξού και έχουμε την σχετική πρόταση για την εισαγωγή αγαθών της πολιτικής κληρονομιάς με παράνομο τρόπο. Προβλέπεται για το πρώτο ε, τρίμηνο του 19 η εξέταση της πρότασης αυτής, αλλά Θα πρέπει βεβαίως να συνοδεύσουμε τις προτάσεις αυτές και με πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εκεί συνεργαζόμαστε με την UNESCO. Κατάρτιση δηλαδή για θέματα αγοράς της τέχνης και προγράμματα κατάρτισης για τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των αστυνομικών δυνάμεων με την παραγωγή ενός εγχειριδίου, τη σύνταξη ενός εγχειριδίου που θα είναι και κάποιων ηλεκτρονικών επίσης εγχειριδίων που θα είναι έτοιμα πολύ σύντομα. Παραλλήλως, ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών και εδώ ο Horizon 2020 μας βοηθάει σχετικά με την προστασία των αγαθών της πολιτικής κληρονομιάς και της ε, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Επίσης διανεγούμε μια μελέτη για την ε, διάσταση του λαθρεμπορίου ε, πολιτιστικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή και των νέων τεχνολογιών που μας βοηθούν στην καταπολέμησή του. Πρέπει να ε, καταλάβουμε περισσότερα για τις οδούς μέσω των οποίων περνάει αυτή, αυτό το παράνομο εμπόριο, της φύσεως και του όγκου των εμπορευομένων των διακινούμενων δηλαδή προϊόντων. Επίσης, στην ευρύτερη σφαίρα της καλύτερης κατανόησης του πότε μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τον κίνδυνο γενικότερος, σε γενικότερο επίπεδο δηλαδή. Έχουμε μια μελέτη και έχω φέρει μαζί μου ένα αντίγραφο αν θέλετε να τη δείτε σχετικά με την προστασία των αγαθών της πολιτικής κληρονομιάς από φυσικές ή τεχνητές καταστροφές και αυτές οι τεχνικές να, να ενσωματωθούν στους ε, τεχνικές της πολιτικής διαχείρισης κινδύνου που έχουν τα κράτη-μέλη αναπτύξει σχετικά με φυσικές και άλλες καταστροφές. Γιατί αυτές μέχρι στιγμής δεν συμπεριλαμβάνουν τα πολιτικά αγαθά. Και προχωρήσαμε λοιπόν σε μια χαρτογράφηση της υφτάμενης πληροφορίας και των πολυάριθμων μελετών που είχαν γίνει στην Ευρώπη. Το σημαντικό πόρισμα που ήδη έχουμε είναι ότι πολύ συχνά δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πολυάριθμες μελέτες και όλες αυτές τις τεχνικές και μελέτες τις χαρτογραφήσαμε σχετικά με το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται στα κράτη-μέλη γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερος και εξού και συνεργαζόμαστε τόσο καλά με την ΓΔΕΛΤΑ ΕΚΟ, το σύστημα πολιτικής προστασίας. Και σε επίπεδο λοιπόν κρατών μελών χρειάζεται να οικοδομήσουμε μια καλύτερη συνεργασία πιο κεντρική πιο ενωσιακή. Και στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντική η δουλειά της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ χρησιμοποιώντας το θαυμάσιο εργαλείο που είναι το σύστημα Κοπέρνικος. Και ο συνάδελφος θα σας το εξηγήσει καλύτερα αργότερα. Τώρα, για την καλύτερη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αγαθών χρειάζεται ένα συντονισμό σε όλα τα επίπεδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικά και περιφερειακά και τοπικά επίπεδα. Γιατί υπάρχει μια έλλειψη ευθυγράμμισης της ε, αλυσίδας αν θέλετε ευθύνης το οποίο σχετίζεται και με το γεγονό ότι ε, ε, η πολιτική κληρονομιά είναι χαμηλής προτεραιότητας αυτή τη στιγμή ή θεωρείται χαμηλής προτεραιότητα. Και βεβαίω έχουμε και την πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών και γνώσεω που αναπτύσσουν οι συνάδελφοι στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Research. Και εδώ έχουμε μια συνολική άποψη όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει για την καλύτερη διαχείριση των πολιτικών αγαθών. και του σχετικού κινδύνου. Δεν θα αναφερθώ περαιτέρω στη διαφάνεια. Άλλο, άλλη σημαντική δουλειά που γίνεται. Είναι τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Γνωρίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε σημαντικές σχολές, σχηματικά κέντρα αριστείας, και σπουδαίους εμπειρογνώμονε. αλλά υπάρχουν διάφορε απειλέ. που αντιμετωπίζει όλη αυτή η εμπειρογνωμοσύνη σήμερα. Αφενός, είναι δύσκολο να διαβιβαστεί η γνώση και η αριστεία μέσω των γενεών. Διότι έχουμε απόσυρση σταδιακή της παλαιότερης γενιάς και αδυναμία μεταλαμπάδευσης αυτής της γνώσης της νεότερη γενία των εμπειρογνωμόνων και οι νεότεροι εμπειρογνώμονες δεν έχουν τα εφόδια που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις διάφορες απειλές. Αν σκεφτούμε ιδιαίτερα την ψηφιακή επανάσταση και το πόσο είναι σημαντικό να διαχειριζόμαστε καλύτερα και με αρτιότητα τα διάφορα ψηφιακά μέσα σχετικά με τις εμπειρίες των επισκεπτών των μουσείων, μεταξύ άλλων, λέει ο Μιλήτρια. Στη Βιέννη λοιπόν πάρα πολύ σύντομα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα πορίσματα αυτής της εξέτασης με συστάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών και για το τι θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλη μια σημαντική πρωτοβουλία, την οποία θα τη διατρέξω σύντομα, λέει η ομιλήτρια, είναι το Heritage for All, για την καλύτερη συμμετοχή και συμμετοχικότητα των τοπικών κοινοτήτων προκειμένου να συνειδητοποιούν την αξία και τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε ένα σημαντικό έργο Άλλη μια πρωτοβουλία είναι το Science for Heritage, με συγχωρείτε. Και εδώ ο συνάδελφος θα σας πει, θα σας δώσει περισσότερα στοιχεία αργότερα. Τα Οι σημαντικές εκδηλώσεις του είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Fair of European Innovators με σημαντική συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων, όχι μόνο ερευνητές, αλλά επαγγελματίες, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, ακαδημαϊκών και μη κτλ. προκειμένου να δούμε πώς καλύτερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σημαντική έρευνα που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να χρησιμοποιηθεί επαρκώς και καταλήλω και από τα κράτη-μέλη. Θα κλείσω με μια προβολή προς το μέλλον. το πρόσφατο θεματολόγιο για, την, για τον πολιτισμό που ενεκρίθη λέει ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την πολιτική κληρονομιά και επομένως τώρα συλλέγουμε όλες αυτές τις εμπειρίες και αντλούμε διδάγματα τα οποία θέλουμε να αποτυπώσουμε σε αυτό το σχέδιο δράση για το μέλλον, γιατί θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε εδώ δεν είναι απλώς σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Τώρα, προφανώς, μια σημαντική συνιστόσα του σχεδίου δράσης θα είναι αυτή η δυνατότητα συνέχισης της προώθησης μιας ολοκληρωμένης και οριζόντιας προσέγγισης για να συνεχίσουμε με ένα σημαντικό και επιτυχέ ε, πρότιμο διακυβέρνηση που θα συμπεριλαμβάνει προφανώ και το επίπεδο των κρατών μελών. Το πρώτο βήμα για μα είναι να συμπεριλάβουμε στον επόμενο διαγωνισμό της Creative Europe παραπομπή στην ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτικής κληρονομιάς ώστε να συνεχίσουμε να ευαισθητοποιούμε σχετικά με τη σημασία του θέματος αυτού και του κοινού αυτού ευρωπαϊκού χώρου. <clears throat> Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας. Θα κλείσω εδώ. Σας ευχαριστώ. Ε, Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στους επόμενους ομιλητές που είναι από άλλες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Θα είδατε ότι η κυρία Σκιακητάνο μίλησε για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βοήθησε στο project αυτό για, την, για το Ευρωπαϊκό Έτος Κληρονομιάς και πρέπει να σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Ε, σύμφωνα με τις συνθήκε, το Κοινοβούλιο δεν δρά ως εκτελεστικός φορέας, εκτελεστική εξουσία. Το Κοινοβούλιο στην περίπτωση αυτή ε, ήταν τμήμα αυτής της, ε, αυτού του project. Οπότε αυτό για μας σήμαινε ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μεγάλη γενοδορία αλλά και κατανόηση από την πλευρά της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της τότε Προεδρίας του Συμβουλίου, της Μαλτέζικης δηλαδή, για την σημασία του, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί η πολιτιστική κληρονομιά σημαίνει μια συλλογή αξιών από όλα τα κράτη. Το γεγονός ότι αυτό το έτος ε, στην, ε, τελειώνει στην ε, Βιέννη, στι στις 6 και 7 Δεκεμβρίου νομίζω ότι είπατε ότι θα γίνει η καταληκτική συνεδρίαση, πάλι αποτελεί ένα σημαντικό συμβολισμό, γιατί αυτή η πόλη, αυτό το κομμάτι του κόσμου δίνει την ουσία της, ευρωπαϊκής, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αποτελεί το, τη γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και πραγματικά αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Ρενέ Μάρτινς από την Γενική Διεύθυνση Έρευνας και την κυρία Γκράσο και τον κύριο Φερκίνη από την ίδια Γενική Διεύθυνση να μας κάνουν τις δικές τους παρουσιάσεις και σας ακούμε. Έχετε το λόγο. Yes, thank you very much. So, Mr. Ευχαριστώ Κύριε Διάκονο, ευχαριστώ που μας καλέσατε σήμερα εδώ σε αυτή την συνεδρίαση. Αγαπητοί εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων και αγαπητοί συνάδελφοι, ε, είναι μεγάλη μου χαρά που μιλώ πάντα εδώ στο Κοινοβούλιο και σας είμαι ευγνώμων. Θα ε, σχολιάσω λίγο ε, αυτά που είπε η συνάδελφος σχετικά με την 7η ε, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία και τους κινδύνους. Κοπέρνικους λοιπόν. Τι είναι ο Κοπέρνικος. Ε, ίσως η παρουσίασή μου να είναι λίγο περίεργη, είναι σύντομη μεν, αλλά θα δείτε δύο πράγματα να συνδέονται που μπορεί να σας φανούν τελείως ασύνδετα. Θα μιλήσουμε για το διάστημα και τι μπορεί να κάνει το διάστημα για την πολιτιστική κληρονομιά. Οπότε το, το παρόν και το μέλλον υποστηρίζει το παρόν και το παρελθόν. Να σα πω δύο πράγματα για το τι κάνουμε. Καταρχά, να σα δώσω ένα γενικό πλαίσιο. Θα γνωρίζετε ίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο ε, διαστημικά προγράμματα. Ένα είναι το Γαλιλαίο για την ευρωπαϊκή ε, πλοήγηση και το GPS και έχουμε και το Κοπέρνικο που ασχολείται με του ε, δορυφόρου που ε, βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη γη για να παρατηρούν τον πλανήτη μα. Και στι δύο περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέχει ουσιαστικά αυτούς τους ε, δορυφόρους, οπότε είναι ένα σημαντικό στοιχείο περιουσιακό σε εισαγωγικά αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μία από τις υποδομές που καμία χώρα ευρωπαϊκή μόνη της δεν θα μπορούσε να έχει. Ο Κοπέρνικος λοιπόν είναι το πρόγραμμα παρατήρησης της ε, γης, είναι το πιο προηγμένο πρόγραμμα, κανένας δεν έχει άλλο τέτοιο πρόγραμμα, ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Μαρικανοί, ούτε οι Ιαπωνέζοι και ε, ολοκληρώθηκε μετά από 20 χρόνια. Οι πρώτες ιδέες για το πρόγραμμα αυτό προτάθηκαν ε, στην Ιταλία, στο Λάγκο Ματζόρε, σε ένα μέρος που ονομάζεται Μπαβένο, πριν από 20 χρόνια. Για να σας πω λοιπόν πώς βελτιώθηκε η παρατήρηση της γης, έχω δύο, δύο φωτογραφίες να σας δείξω που δείχνουν το σημείο ακριβώς αυτό που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία. Εδώ βλέπετε την φωτογραφία της Λάγκο Ματζόρε πριν από 20 χρόνια που ελήφθη από έναν Αμερικανό, αμερικανικό δορυφόρο, τον Landsat. Εδώ βλέπετε το ίδιο σημείο με φωτογραφία που ε, βγήκε από τον Ευρωπαϊκό Δορυφόρο, τον Sentinel-2, στις 14 Ιουνίου του 2018. Βλέπετε λοιπόν πόσο τεράστια είναι η διαφορά α, στην... Α, καθαρότητα της, στην ευκρίνεια της ε, εικόνας και μπορούσα, θα μπορούσα βέβαια να σας πω πολλά για το τι κάνει άλλα ο Κοπέρνικος αλλά ε, νομίζω ότι βλέπετε πραγματικά εδώ τι κάνουμε. Έχουμε λοιπόν τους δορυφόρους βλέπετε στο κέντρο της διαφάνειας. Και χάρη στα δεδομένα που έχουμε και τις απεικονίσεις από αυτούς τους δορυφόρους, μπορούμε να έχουμε πληροφορίες από διάφορους τομείς. Μπορούμε ας πούμε, να παρατηρήσουμε τα θέματα της γης, του ατμοσφαιρικού αέρα, της θάλασσας, Μπορούμε να υποστηρίξουμε επίγουσες δραστηριότητες πολιτικής προστασίας, για παράδειγμα, ε, δραστηριότητες ασφάλεια, μέσω ασφάλειας της θάλασσας, ε, αντιμετώπιση της ε, πειρατεία, του λαθρεμπορίου, κλιματική αλλαγή επίσης. Παρατηρούμε μέσω των δορυφόρων πώ λιώνουν σιγά σιγά οι πάγοι στους πόλους. Τώρα, πώς συνδέονται όλα αυτά με την πολιτιστική κληρονομιά. Όταν μιλούμε για πολιτιστική κληρονομιά, εδώ βλέπετε την ε, διαφάνεια που, έχουμε, ε, που είχαμε σε ένα από τα εργαστήρια για την ε, πολιτιστική κληρονομιά και το διάστημα, βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα, πολλές, πάρα πολλοί χώροι που θεωρούνται πολιτιστική κληρονομιά. Ε, τα στοιχεία αυτά είναι από την UNESCO βέβαια, δεν θα είναι τα τελευταία, μπορώ να σας δώσω και άλλα στοιχεία αν θέλετε και βλέπετε ότι έχουμε πολιτιστικούς στόπους ε, και είναι πάρα πολλά σημεία αυτά τα οποία μπορούμε τελικώς να παρατηρήσουμε. Εδώ βλέπετε εικόνες που μπορεί να πάρει κανείς από το δορυφόρο. Ο δορυφόρος πετάει περίπου στα ε, χίλια χιλιόμετρα πάνω από τη γη. Λαμβάνοντα υπόψη ότι ένα αεροπλάνο πηγαίνει γύρω στα 10 με 12 χιλιόμετρα, σημαίνει 100 φορέ παραπάνω. Άρα έχουμε αυτή και καλύτερη ακόμη απεικόνηση, οπότε οι, δορυφόροι μπορούν να, πάνε, να φτάσουν μέχρι απεικόνηση 30 εκατοστά από τη γη. Ε, Βεβαίω ε, αυτές οι φωτογραφίες είναι από το ίντερνετ, έχουμε και εμεί δικές μας, αλλά εδώ βλέπετε την Αίγυπτο, την Αυστραλία, η τρίτη είναι η Σαμάρα στο Ιράκ, ε, το Αγκόρ, η, η μεσαία είναι ο καρολογινή ύφαλο στην Αυστραλία και η τελευταία είναι μια μυστική, ξεχασμένη πόλη στη Σαχάρα που καταγράφηκε μέσω παρατήρησης από το δορυφόρο. Ποιες είναι τώρα οι απειλές στην πολιτιστική κληρονομιά. Καταρχάς, να δούμε τι κάνει η ατμοσφαιρική ρήπανση στην πολιτική κληρονομιά, η οποία μπορεί πραγματικά να επιτεθεί στους χώρους κληρονομιάς. Το δεύτερον, πόλεμος, βομβαρδισμοί μπορεί να καταστρέψουν χώρου ε, χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν υπάρχει κανένας τρόπος αυτό να σταματήσει. Τρίτος λόγος, φυσικές καταστροφές σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, που σιγά σιγά εξαφανίζονται, Πλημμύρε, αποψήλωση δασών, σεισμοί. Αυτά είναι πραγματικά ε, ε, κίνδυνοι που επιτίθενται στις, ε, στους χώρους πολιτικής χρονομιάς και αυτό που μπορούμε να κάνουμε μέσω του Κοπέρνικους μπορεί όντως να βοηθήσει γιατί μπορούμε να αναλύσουμε ας πούμε την ποιότητα του αέρα και να δούμε ποια είναι τα επιβλαβή στοιχεία και να βελτιστοποιήσουμε την παρέμβασή μας σε χώρους πολιτικής χρονομιάς που πλήττονται από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Επίσης μπορούμε να συγκρίνουμε τι έγινε πριν και μετά από μια επίθεση, μετά από ένα βομβαρδισμό, να δούμε ποιε είναι οι περιοχέ που καταστράφηκαν για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε την καταστροφή και να βοηθήσουμε να καταγραφούν οι ε, παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Επίσης, για τις φυσικές καταστροφές μπορούμε να προβλέψουμε ε, ε, κινδύνους για τους τουρίστες που επισκέφτονται την περιοχή και να αλλάξουν, για να τους προετοιμάσουμε να αλλάξουν το, το, τα μέρη που θα επισκεφθούν. Επίσης, πολιτική προστασία, να δούμε ποιες είναι οι περιοχές που πλήττονται σημαντικά από ψήλωση. Ξέρετε τι γίνεται. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικός κίνδυνος, μειώνονται δάση που έχουμε σε όλη την ε, σε όλο τον πλανήτη. Μπορούμε κάθε χρόνο, κάθε μήνα ακόμη να υπολογίσουμε πόση, πόσο της εκατό των δασών αποψηλώνεται και επίσης οι, α, σεισμοί. Μπορούμε να καταγράψουμε που γίνονται, μπορούμε να καταγράψουμε ποια είναι η ζημιά που γίνεται και ποιο κομμάτι του χώρου πολιτιστικής κληρονομιάς έχει α, καταστραφεί. Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε χάρτες που θα περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη με το κέντρο της Ρώμης. Μέσω συγκεκριμένων τεχνικών μπορεί κανείς να ε, δει πώς κινείται η γη. Ε, κάποιες περιοχές ε, κινούνται προς τα πάνω, κάποιες βυθίζονται, οπότε αυτό μπορούμε να το ενσωματώσουμε στα στοιχεία που έχουμε και έτσι μπορούμε να προβλέψουμε κάποιες παρεμβάσεις ή να προγραμματίσουμε κάποια μεγαλύτερη υποπτία για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Εδώ βλέπετε στη Συρία προσπαθήσαμε να δούμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στην περιοχή. Η φωτογραφία που βλέπετε στο τέλος είναι υψηλή ε, ευκρίνειας από το Google Earth. Έχουμε ε, και κάποια, από το Sentinel έχουμε κάποιες ε, φωτογραφίες μικρότερης ευκρίνειας, αλλά μπορούμε να έχουμε μια νέα εικόνα κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 3-4 χρόνια. Έχουμε μια διάμετρο 10 μέτρων αλλά βεβαίω δεν μπορεί πονή, ποτέ κανεί να βγάλει φωτογραφία κάθε δύο-τρει μέρε. Πάνω, πάνω πάνω στις φωτογραφίες μπορούμε να καταγράψουμε τις αλλαγές που γίνονται στο πολιστικό αυτό μνημείο. Ε, βλέπουμε ποια είναι η κατασκευή που έγινε από τις 4 μέχρι τις 18 του 2016. Και τούτων λεχθέντων ήδη Σήμερα έχουμε τις υπηρεσίες του Κοπέρνικος που ελέγχουν τον αέρα, την κίνηση των εδαφών και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε. Ας πούμε για, τις, για τους σεισμούς, για την μετακίνηση των γεών. Ή μπορούμε να ελέγξουμε την μόλυνση, μπορούμε να βρούμε θαμένους πολιτικούς χώρους, καταστροφή, κλιματική αλλαγή, χρήση των γεών και πώς αυτή αλλάζει. Όλα αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τις παρεμβάσεις μας. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Τι μπορούμε να κάνουμε για την στήριξη της ε, πολιτικής κληρονομιάς. Υπάρχει μια task force η οποία ελέγχει το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το προϊόν που έχουμε για την πολιτική κληρονομιά, τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή Κοπέρνικου συμφώνησαν να διερευνήσουν πώς μπορεί να γίνει αυτό. Η Ιταλία προσφέρθηκε να πάρει τον ηγετικό ρόλο και υπάρχουν αρκετά που έχουν συμπεριληφθεί στην Task Force που ξεκινά την εργασία τη αυτές τις ημέρε. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι καμιά φορά αυτοί ε, οι, δορυφόροι είναι μόνο για ειδικού. Το θέμα είναι ότι είναι καλά στοιχεία αυτά και για τους ε, χρήστες, γιατί μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους ώστε οι τελικοί χρήστες να ξέρουν τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο ένας δορυφόρος. Και επίσης υπάρχουν ε, και ε, εγκύκλοι στα πανεπιστήμια για την, και στην ανώτερη εκπαίδευση για, με το θέμα αυτό, που χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά των δορυφόρων. Αυτά έτσι συντόμως από μένα, εισαγωγικά. Αν θέλετε περισσότερες ε, πληροφορίες υπάρχει η σελίδα μας, εκεί μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε και βεβαίως αν υπάρχουν ερωτήσεις ευχαριστώ να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε... Χαίρομαι που είμαι εδώ να σας παρουσιάσω τι κάνουμε για να στηρίξουμε την επιστήμη σχετικά με την πολιτική κληρονομιά. Θα σας μιλήσω για την πρωτοβουλία 10. Ε, σας θυμάστε, σας παρουσίασε τις 10 ε, πρωτοβουλίες συναδελφός μου. Ε, τι είναι η διατήρηση πολιτικής κληρονομιάς. Θέλω να χρησιμοποιήσω την εξή αναλογία. Ξέρουμε τι κάνει ένας γιατρός, τι είναι η πρόληψη, τι είναι η θεραπεία. Το αντίστοιχο στην πολιτική κληρονομιά είναι ότι η ίδια πολιτική κληρονομιά είναι ο ασθενής, ο συντηρητής είναι ο γιατρός που χρησιμοποιεί τις, τη γνώση του για να αποφασίσει ποια θα πρέπει να είναι η θεραπεία. Ε, τα φάρμακα είναι οι ουσίες που χρησιμοποιούνται, τα υλικά που χρησιμοποιούνται και η εγχείρηση ε, έχει το αντίστοιχό της ε, στην ε, παρεμβατική συντήρηση. Και βέβαια έχουμε και την πρόληψη, όπως και στην ανθρώπινη υγεία, έχουμε πρόληψη και στην πολιτική δεν την αγγίζουμε την πολιτική κληρονομιά, παίρνουμε μέτρα έτσι ώστε να μην ζημιωθεί, να μην βλαφθεί. Επίσης χρειάζονται και στις δύο περιπτώσεις υψηλά και αυστηρά ε, ψηλές και αυστηρές προδιαγραφές, ε, δεοντολογικές προδιαγραφές. Ο ασθενής, ε, από την άλλη μεριά, είναι ένα άτομο και το κάθε άτομο έχει τη δική του ανάγκη διάγνωση. Έτσι αυτό ισχύει και για κάθε στοιχείο της πολιτικής κληρονομιάς. Η πολιτική κληρονομιά είναι τμήμα των προγραμμάτων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1996 και του Horizon 2020. Το Horizon 2020 αφιέρωσε περίπου μισό δισεκατομμύρια ευρώ στην πολιτική χρονομιά. Αυτό αποτελεί μια αύξηση σχεδόν 100% σε σχέση με το προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το, ε, ε, ε, το, η συνάδελφός μου στο πάνελ 1 θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, θα τα δείτε γραπτά για τα ποσά που χρησιμοποιούνται αυτά τα ποσά στις ε, τεχνικές ε, για την πολιτική χρονομιά. Ε, το πρόγραμμα NMBP αφορά τις νεοτεχνολογίες, ε, τα σύγχρονα υλικά, βιοτεχνολογία και τις τεχνικές. Σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας καλύπτουμε συστηματικά προληπτικές μεθόδους χαμηλού κόστους αλλά και συγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης νέων υλικών και λύσεων. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το ε, τέλος του 2020, πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ, οκταπλάσια δηλαδή ποσά για αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με το προηγούμενο, το έβδομο πρόγραμμα. Έχουμε βέβαια και άλλα προγράμματα. Ε, γι' αυτό το λόγο ο συνολικό προπολογισμό είναι μεγαλύτερος. Αυτό το πρόγραμμα όμως παίρνει 45 εκατομμύρια ευρώ. Να σας δώσω μερικές εικόνες από πρόσφατα project που είτε ολοκληρώθηκαν είτε συνεχίζονται στο πλαίσιο του Horizon 2020. Έχουμε τον καθεδρικό αυτό με προστατευτικά υλικά για διάφορες λιθοδομές. Αυτά χρησιμοποιούνται συχνά σε τέτοιου είδους ε, παλιούς ναούς, αλλά και για την όπερα του Όσλο πολύ διαφορετικό κτίριο, πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο. Δύο διαφορετικά κτίρια λοιπόν που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνική. Η Innova Concrete ε, χρησιμοποιεί οι τεχνικές για να προστατευθούν ε, κτίρια που είναι χτισμένα από μπετόν. Από την Πολωνία, από την Ισπανία, βλέπετε διάφορα παραδείγματα εδώ. Το επόμενο, η επόμενη διαφάνεια είναι ένα project που ασχολείται με την προστασία ε, πολιτικής ε, σε μορφή σελουλόιντ, ε, φιλμ, κινηματογραφικά φιλμ, ταινίες κλπ. Το Nano Restart ε, αφορά νέες τεχνικές και υλικά για την διατήρηση ζωγραφικών πινάκων. Εδώ βλέπετε του Πόλου και του Πικάσο δύο πίνακες. Για όλα αυτά ε, είναι πολύ σημαντικά τα επιτεύγματα, τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε δηλαδή από την κοινότητα των συντηρητών τέχνης, των επιστημόνων κλπ. είναι πολύ θετικά. Και τι λένε αυτά τα μηνύματα, λένε ότι η επιστήμη για την πολιτική κληρονομιά υποχρηματοδοτείται πάρα πολύ. Ε, η χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο είναι, η χρηματοδότηση είναι χαμηλή και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είναι μια ανησυχία και ε, ένα πρόβλημα το οποίο μας το αναφέρουν συχνά θα πρέπει να αυξηθούν τα ποσά τα οποία χρηματοδοτούν επιστημονικές έρευνες για θέματα πολιτικής κληρονομιάς. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές, σημαντικές πρόοδοι στην ψηφιοποίηση της πολιτικής κληρονομιάς, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Ε, αυτή η εργασία βοηθάει προφανώς τη συντήρηση των εργοτέχνης, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα ίδια τα έργα τέχνης, τα ίδια τα έργα της πολιτικής κληρονομιάς. Ε, η ψηφιοποίηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη διάφορες πτυχές, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική κλπ. Αλλά και διοικητικές πτυχές, όπως για παράδειγμα οι δημόσιοι διαγωνισμοί πολύ συχνά θεωρούν ότι η συντήρηση αποτελεί μια απλή εφαρμογή υπαρχουσών τεχνικών. Ε, η έρευνα είναι, θεωρείται πολύ περιορισμένη, όμως ε, στην συντήρηση και ε, ε, ανάταξη ενό έργου τέχνη, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που χρειάζονται σημαντική έρευνα για να βρεθεί μια λύση. Επίση, χρειάζονται βέλτιστες πρακτικέ και διεθνή πρότυπα. Αυτό μα το αναφέρει η κοινότητα. Κάποιε χώρε έχουν σημειώσει πρόοδο και στι προδιαγραφέ και στι διαδικασίε. Αυτέ οι βέλτιστες πρακτικέ, αυτά τα βέλτιστα στάνταρ θα πρέπει να γίνουν και ευρωπαϊκά. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ίσως κάποιες ε, ερωταπαντήσεις τώρα. Θα σας ε, ζητούσα να περιοριστείτε στα δύο λεπτά στις ερωτήσεις σας ε, και να κάνετε μια σύντομη εισαγωγή προτού ρωτήσετε. Και μία παρατήρηση από πλευρά μου, αν ε, μπορώ. Αυτή είναι η τελευταία μορφή δικτατορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το σφυράκι εδώ που κρατάω, και θα λειτουργήσει, λέει ο Πρόεδρος. Διότι όλοι εδώ έχουμε τρόμο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ενός λεπτού, γνωρίζετε την πίεση αυτή όλοι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μετά από μια σύντομη παρουσίαση Παρακαλώ, τις ερωτήσεις σας. Καλημέρα σας. Στις 6 ε, και 7 Δεκεμβρίου θα γίνει στη Βιέννη η καταληκτική συνεδρίαση και χαιρόμαστε που μπορούμε σήμερα να παρουσιάσουμε αυτό το, αυτή την εκδήλωση και σήμερα. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον χρόνο που μου, που μου δώσατε για να σας ε, αναφέρω κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες υπάρχουν ε, για το πώς, για το τι γίνεται στον τομέα της πολιτικής κληρονομιάς. Ε, έχουμε την UNESCO η οποία ασχολείται βεβαίω με την πολιτιστική κληρονομιά και με τα διάφορα project, γιατί υπάρχουν κάποια προγράμματα για την δημιουργία ουρανοξύστης στα κέντρα της πόλης. Στις, είναι κρίμα που σε αυτή την ε, σημερινή συγκυρία αυτό δεν έχει ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη. Βεβαίως αυτό υπουργείο, τέτοιο υπουργείο στην Αυστρία δεν υπάρχει πολιτιστική κληρονομιά. Είναι πάντα περιφερειακό ή τοπικό το, η αρμοδιότητα αυτή. Και βεβαίω αυτό σημαίνει ότι οι ε, ε, τιμές των ε, κτίριων αυξάνονται λόγω ακριβώς των νέων κατασκευών. Ε, οπότε νομίζω ότι αυτή είναι λίγο αμφίροπη ε, συμπεριφορά απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά. Η πολιτική δεν παρεμβαίνει αποτελεσματικά για να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά. Και αυτό το θέμα δεν είναι θέμα βιωσιμότητας ή κοινωνικής ε, ατζέντα. Είναι ένα θέμα στο το οποίο προωθεί πάρα πολύ το λόμπι των κατασκευαστών, κατασκευαστικών εταιριών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω για τη διατήρηση της ε, πολιτικής κληρονομιάς ε, να κοιτάξετε και λίγο πίσω από τις ε, λέξεις και να προστατεύσετε το, την πολιτική κληρονομιά στην Βιέννη από τέτοιες πρακτικές. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, Φελίθ Μόντες, γερουσιαστής από την Ισπανία. άκουσα τις εξηγήσεις που μας δώσατε για την πορεία από το 2014 στο 2018 μαζί με αυτό το ευρωπαϊκό έτος για την πολιτιστική κληρονομιά. Επί τη βάση των πρωτοβουλίων αυτών είχαμε τους πυλώνες που μας ε, παρουσιάσατε. Τώρα η προώθηση και η υποστήριξη που θέλουμε να δώσουμε στην πολιτική αυτή θα έπρεπε να αποτυπώνει και άλλους πυλώνες που είναι θεμελιώδεις για την ε, ενωσιακή δομή και αυτό να το εκφράσουμε ρητά την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και εδώ επιτρέψτε μου ως πρώην από την περιφέρεια της Σεγόβια να σας ε, μιλήσω για την πολιτιστική κληρονομιά της υπαίθρου που είναι πάρα πολύ σημαντική για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλληλεγγύη λοιπόν. Άλλη σημαντική αρχή και πυλώνας θα ήταν η κοινωνική ισότητα, δικαιοσύνη, εργασιακή, οικονομική και κοινωνική. Δεν μπορούμε να μιλούμε για βιώσιμο τουρισμό αν δεν αναφερόμαστε επίσης στα θέματα εργασιακού δικαίου και ισότητας. Τρίτο στοιχείο θα ήταν η προσβασιμότητα και για τους δημιουργούς και για το κοινό. Και ε, τέλος, σημαντικός επίσης πυλώνας είναι η συμμετοχή στα συστήματα και προγράμματα παιδείας και ε, ε, η διαβίβαση αυτών των αξιών και αρχών οριζόντια και για να μην μακρηγόρησε ο Πρόεδρε, το σημαντικό από αυτά που ακούσαμε εδώ είναι ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτήν την έννοια των πολιτικών για τον πολιτισμό και να μιλήσουμε για, ένα, για μια ευρύτερη έννοια που θα αφορά σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια για την προστασία ως δικαίωμα, θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά και πόρο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα εκπρόσωπος του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις παρουσιάσεις σας. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω. Ζητούν από την ομιλήτρια να μιλάει πιο κοντά στο μικρόφωνο. Πράγματι δεν ακουγόταν. Ζητώ συγγνώμη λέει ομιλήτρια. Αναφέρθηκα λοιπόν στις παρουσιάσεις. Είναι κάτι που θα ήθελα να σημειώσω από αυτά που είπε η εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν για τις φυσικές και άλλες καταστροφές το οποίο δεν συνηθίζεται ίσως σε νοσιακό επίπεδο, αλλά στην Ισπανία είχαμε τέτοιες ε, εμπειρίες όπως σε συγκεκριμένους σεισμούς κοντά σε πολιτικά κέντρα. Και επομένω, υπό την έννοια αυτή η προστασία της πολιτικής οικονομίας δυσκολεύεται από την έλλειψη ειδικών εμπειρογνωμόνων, ειδικών, τεχνικών που να εργάζονται σε συγκεκριμένα κέντρα και για τα προγράμματα της κατάρτισής της για την αποθήκευση, για τις ε, τεχνικές αποκατάστασης ε, συγκεκριμένων μνημείων και αυτά χάνονται σιγά σιγά και προκειμένου να προστατεύσουμε το σύνολο της κληρονομιάς δεν είναι δυνατόν πάρα πολύ συχνά αν δεν έχουμε τεχνικούς που να έχουν την ειδίκευση που απαιτείται και τη γνώση που απαιτείται. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για την προστασία συνολικά της πολιτικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φεντερόβιτς ε, γυριστή από την Πολωνία ασχολούμαι τα θέματα πολιτισμού ε, στην ε, Πολωνική Γερουσία και θα ήθελα να πω στην συνάδελφο από την Ισπανία ότι για, σχετικά με την αποκατάσταση έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα ε, κατάρτισης. Συνεργαζόμαστε και με γειτονικές χώρες. Θα μιλήσω και αύριο για τις επαφές που είχαμε με την Ουκρανία γιατί έχω προγραμματισμένη παρέμβαση αύριο, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα φάκελο όπου μιλούμε για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας ε, της Βαρσοβίας. Είχαμε και μία συνάντηση με άνω των 200 συμμετεχόντων, όπου παρουσιάστηκαν συστάσεις πάρα πολύ σημαντικές και θα ήθελα να το αφήσω αυτόν τον οδηγό στη διάθεση των συναδέλφων, των μελών, ε, γιατί είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι συστάσεις, διατίθενται και στο διαδίκτυο. Ίσως μιλούμε για κάτι ε, λιγάκι προφανές. Εγώ χρόνια ε, τώρα ασχολούμαι με τα θέματα προστασίας ε, του πολιτισμού. Είχαμε αναπτύξει και ένα κώδικα στην Βαρκελόνη, με το 2003, και ως προς αυτό διανύουμε ένα σημαντικό σημείο καμπής στην ιστορία της Ευρώπης ε, και είναι χάρη στον πολιτισμό και στην παιδεία που μπορούμε σήμερα να ε, ε, πείθουμε τους πολίτες να μας εμπιστεύονται και να ακολουθούν αυτές τις αρχές και τις αξίες που προσπαθούμε να προασπιστούμε. Και αναφερόμαστε σε διεθνή σώματα, φορείς στην UNESCO, στην ε, Παγκόσμια Τράπεζα, σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την προστασία της πολιτιστικής κλονιάς. Θα το δώσω αυτόν τον οδηγό στον πρόεδρο για να τον διαβάσουν όλοι οι συνάδελφοι όσοι ενδιαφέρονται. Παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος. Ε, ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Ένα ερώτημα ακόμα Α, ένα ερώτημα ακόμα θα επιτρέψουμε και μετά να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές για να απαντήσουν. Σας ακούμε. Ε, είμαι Δημήτρης Σεβαστάκης από το, κοινοβούλιο, το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ε, το ερώτημά μου ξεκινάει από, αυτό που, από την παρατήρηση της συναδέλφου για τη βιωσιμότητα. Υπάρχει ένα πρόβλημα ιδεολογικής βιωσιμότητας, όχι μόνο οικονομικής. Η το έβριμα, το πολιτιστικό, διασταυρώνεται με πολεοδομικά, χωροταξικά, προβλήματα ανάπτυξης, αγροτικής οικονομίας, παραγωγής, μόλυνσης, όλα αυτά που αναφέρθηκαν. Υπάρχει μια, ένα αργό δίκαιο που προσαρμόζεται σε αυτό το ε, δυσεπίλητο πρόβλημα που είναι ανάπτυξη, που είναι αναπτυξιακό, αλλά και κυρίως αφορά την πολιτιστική αφομοίωση του ε, κληροδοτήματος από τη σύγχρονη ζωή. Ε, η ανάπτυξη της πόλης, η ανάπτυξη των αναγκών και κυρίως μια παιδεία εικονογραφική ε, που οδηγεί όχι πια στο έβριμα, αλλά στην αφήγηση γύρω από το έβριμα, μέσα από τα animation, μέσα από το παραστατικό μουσείο που συστήνεται, αυτό σαν πρόβλημα δημιουργεί, κατά την προσωπική μου γνώμη, και θέτει ένα ερώτημα ιδεολογικής βιωσιμότητας ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και γι' αυτό ε, σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να θεσμίσει όρους νομικής και τεχνικής προστασίας του ε, ευρήματος, του κληροδοτήματος. Merci. Merci. Ε, σας ακούμε. Λιλιάνα Σπούνα, είστε νούμερο με σενατόρ. Λιλιάνα Σπούν ονομάζομαι. Είμαι ε, γερουσιαστής στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο και είμαι μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης. Ε, χάρηκα πολύ μετά όσα άκουσα από τις ε, παρουσιάσεις, κυρίως ό,τι αφορά την ε, σύγκριση μεταξύ ιατρικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Μου άρεσε πολύ. Η πολιτιστική κληρονομιά φαίνεται να πάσχει αυτή τη στιγμή, αν δούμε αυτή τη σύγκριση που κάνατε. Στην ε, Ρουμανία οι γιατροί δυστυχώς μεταναστεύουν σε άλλες χώρες. Και ακόμα και αν ε, έχουμε όλο και περισσότερε θέσει εργασία για γιατρού, ακόμη και αν είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, αν προετοιμάζουμε του φοιτητέ μα και τα πανεπιστήμια, δυστυχώ οι γιατροί φεύγουν από τη χώρα μα και με την εθνική, ε, μετά από τα πάθη της ε, ιατρικής υπάρχουν και τα πάθη της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τα διαρθρωτικά ταμεία για την πολιτιστική κληρονομιά τα οποία βεβαίω είναι πάρα πολύ χρήσιμα στη Ρουμανία και με τη βοήθεια των διαρθρωτικών ταμείων έχουμε καταφέρει να κάνουμε πολλέ αποκαταστάσει πολιτιστικών μνημείων, αλλά υπάρχουν βεβαίω πολλέ προποθέσει οι οποίε μα δυσκολεύουν την πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια. Μία εκ των οποίων είναι ότι μετά την αποκατάσταση, μετά την ανακαίνιση, το, ε, το κτίριο πρέπει να είναι προσβάσιμο από το κοινό. Αλλά το κτίριο αυτό Συνήθω είναι κάποιο κτίριο στο οποίο στεγάζεται κάποιο δημαρχείο ή κάποια δημόσια υπηρεσία. Μπορεί μόνο να επιτρέψει την πρόσβαση μόνο σε ένα κομμάτι, στο κοινό, σε ένα κομμάτι του κτίριου μόνο αυτού. Οπότε, ίσως θα πρέπει οι κανόνες αυτοί και των διαρθρωτικών ταμείων να αλλάξουν για να μπορέσουμε κι εμεί να ανακαινίζουμε περισσότερα κτίρια. Μιλήσατε για τον τρίτο πυλώνα και την προστασία για τα ποιοτικά συστήματα, για τον έλεγχο της ε, ποιότητας, για το, καθ' όλη τη διάρκεια της ε, ζωής ε, του προγράμματος αυτού, έλεγχοι δηλαδή που θα λειτουργούν και μακροπρόθεσμα, αλλά αν δούμε τις συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες θα μπορεί κάθε χώρα να παίρνει μέρος, τότε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι χώρες ε, για να μπορούν ε, όλες να συμμετάσχουν, να συμμετάσχουν στην ε, εκπόνηση των κριτηρίων. Λοιπόν, σύντομα παρακαλώ τις παρεμβάσεις σας, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε χρόνο να απαντήσουν. Προηγούμενους ομιλητές για τις πολύτιμες εισηγήσεις, τις οποίες έχουν παραθέσει. Ταυτόχρονα όμως να, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη πέραν από την προστασία και τις και της πολιτικής της καταγραφής και της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι κίνδυνοι οι οποίοι, και οι επιθέσεις οι οποίες ε, δέχεται η πολιτιστική κληρονομιά είναι τόσο μεγάλη και επικοιλόμορφοι. Δεν αναφέρομαι μόνο στους κινδύνους α, ε, στις περιοχές κρίσεων ή στις περιοχές όπως στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου ή ακόμη και αυτά τα οποία έχουμε ζήσει στην Συρία και το Ιράκ, όπου με μιας έχουν αφανιστεί από το χάρτη κάποιες α, ε, α, ε, πολιτιστικές ε, ιδιοκτησίες, αλλά και από το περιβάλλον. Έχουμε κινδύνους τέτοιους, οι οποίοι με μιας μπορούν να αφανίσουν τέτοιου είδους πολιτιστικές ιδιοκτησίες. Θέλω με αυτό, με αυτό το, να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ είναι που μπορούμε να εσκύψουμε, μέσω της ψηφιοποίησης να ενδυναμώσουμε την αρχή της καταγραφής. Όλα αυτά μπορούν, να καταγραφούν. Όλα αυτά μπορούν να αποτυπωθούν ηλεκτρονικά, ούτω ώστε να υπάρχει και ευχέρεια μετά από την οποιανδήποτε εξέλιξη ή κίνδυνο ή καταστροφή, στη συνέχεια να υπάρχει η δυνατότητα της αποκατάστασης ή της επαναφοράς στις, στην αρχική τη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λέει ο πρόεδρο, ε, θα ζητούσα τώρα από του ομιλητέ μα. Ε, Ποιο θα ήθελε να απαντήσει. Ο κύριο ε, Φακή. Βεβαίως, να απαντήσω εγώ, Πρόεδρε, μερικώς, λέει η κυρία Σακίνο. Βεβαίως και έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αναλάβουμε δράσεις σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τώρα, ε, αρκετές από τις ερωτήσεις σας επιβεβαιώνουν την ανάγκη πιο ολιστικής προσέγγισης στο ζήτημα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πίεση της ανάπτυξης αν δεν συνεργαστούμε καλά, επί παραδείγματι, για την καλύτερη ενημέρωση και κατάρτιση του κοινού για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί αυτό εν είδη μέσω συνένεσης δηλαδή της κοινή νόμης μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται δηλαδή την πραγματική αξία Επίσης η απαγόρευση πρόσβασης του κοινού σε συγκεκριμένους χώρους και εδώ αναφέρομαι στο θέμα της προσβασιμότητας, εάν δεν μπορούν να απολαύσουν τους χώρους και τα μνημεία αυτά, πώς να αντιληφθούν την αξία του και επομένως προσβασιμότητα είναι πρώτο και σημαντικότατο στοιχείο. Ε, στις 4 Δεκεμβρίου να επιβεβαιώσω ότι θα απονείμουμε το Access City Award που είναι βράβευση από πλευρά τη Επιτροπής προ τα αστικά εκείνα κέντρα που προσπαθούν να καταστούν πιο προσβάσιμα για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Στα μνημεία δηλαδή πολιτιστικής κληρονομιάς. Και για πρώτη φορά δεν έχουμε μόνο μία βράβευση για πόλεις άνω των 15.000 κατοίκων, αλλά και συγκεκριμένη βράβευση για τις πιο μικρές. Και ακριβώς εδώ προσπαθούμε να υπογραμμίσουμε την σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κέντρα της Υπέθρου 4 Δεκεμβρίου θα είναι η τελετή αυτή, η απονομή αυτή, που είναι η μέρα των ανθρώπων με αναπηρία. Ε, και πάλι, πρέπει να εργαστούμε στα θέματα της κατάρτισης και εκπαίδευσης των ε, ειδικών, των επαγγελματιών, συμφωνώ πολύ τους δηλαδή, έχουμε επεξεργαστεί συστάσεις ε, από πλευρά της ομάδας εμπειρογνωμόνων, με εμπειρογνώμονες και από το πεδίο, από την παιδεία και από τον πιο συγκεκριμένο χώρο του πολιτισμού, γιατί βεβαίως έχουμε ένα ευρωπαϊκό πεδίο, ε, με συγχωρείτε, πλαίσιο για, τον, ε, για την παιδεία και αναφερθήκατε και στις στους ε, επαγγελματίες, ε, στους ειδικού ε, σε θέματα αποκατάστασης. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ακαταρτισμένους τεχνικούς, δεξιοτέχνες που να ασχολούνται με αυτά τα θέματα με προγράμματα κύκλου ζωής και τα οποία να εξασφαλίζουν ότι θα διαβιβάζεται πράγματι αυτή η γνώση, όπως έλεγα και νωρίτερα, στους νεότερους τεχνικούς. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια ορολογιακή βόμβα. Πρέπει να προλάβουμε η γνώση αυτή να διαβιβαστεί από αυτούς που απέρχονται, που αποσύρονται, που συνταξιοτούνται δηλαδή αυτή τη στιγμή, προς τους νεότερους Ε, αυτά θα έλεγα από πλευρά μου. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων, δεν είμαι ειδικό, δεν θα ήθελα να θεωρήσω ότι είμαι σε τεχνικά δηλαδή σε θέση να δώσω απαντήσεις εδώ, αλλά αναφερθήκαμε συχνά σε ε, κάποιο είδος ε, κινδύνου στρατιωτικών παρεμβάσεων σε κάποια μέρη του κόσμου και περιβαλλοντικών κινδύνων, αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια βραδία βία που ασκείται άλλου είδους και θα την ονόμαζα εμπορική, αγορέα βία. Δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο διεισδύει η αγορά ή στην περιοχή του πολιτισμού, γιατί έχουμε αγαθά ε, που έχουν καταστραφεί απολύτως ε, λόγω οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων. Δηλαδή στοιχεία κτηρίων που επικαλύφθηκαν από τσιμέντο, τέτοιες λεπτομέρειες. Και αυτό οφείλεται σε άγνοια, άγνοια. Και άγνοια τεχνικών, άρτιων τεχνικών αποκατάστασης ε, κτηρίων και μνημείων. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε νομίζω στο δεύτερο γύρο με τον κύριο Παπούλια της ε, ΓΔΕΝΒ, ο οποίος θα έχει τώρα το λόγο για την δική του παρουσίαση, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε στη συνεδρίαση. Εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος στην ε, μονάδα που ασχολείται με την προστασία της φύσης και θα ήθελα να σα ε, κάνω μια γενική παρουσίαση των ε, δραστηριοτήτων της Γενική Διεύθυνση για να μπορέσουμε να διαρευνήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ της φυσικής και της πολιτισμικής κληρονομία. Το επίκεντρο της δουλειάς μας είναι οι ευκαιρίες που μας ε, δίνονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις προστατευόμενες περιοχές, το Natura 2000, το οποίο, όπως ξέρετε, είναι ο πυλώνας της πολιτικής για τη βιοπικιλότητα και στόχο έχει να διαχειρίζεται ε, και να ε, αποκαθιστά τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα και τα πιο ευαίσθητα είδη στην Ευρώπη. Το δίκτυο αυτό καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι της επικράτειας των κρατών μελών και διευρύνεται και στη θάλασσα. Οι σχέσεις τώρα των προστατευόμενων περιοχών για στόχους ε, διατήρησης της ε, φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει μπει σε τα τελευταία χρο... Έχουν μπει σε συζήτηση τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν ε, αρκετοί σημαντικοί λόγοι γι' αυτό. Καταρχάς διότι πολλά από τα προστατευόμενα οικοσυστήματα σχετίζονται και με πολιτιστικά σημεία, με πολιτιστικούς τόπους που είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς ε, των ε, ανθρώπων τις τελευταίες εκατοντάδες χρόνια. Ε, υπάρχει λοιπόν σημαντική σχέση μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητα και της φύσης. Και επίσης το γεγονός ότι έχουμε πολύ σημαντικές επικαλύψεις χωροταξικές μεταξύ ε, ε, χωρών προστατευόμενων αλλά και με χώρους που έχουν σημαντική πολιτιστική σημασία, αρχαιολογικούς χώρους ας πούμε ή χώρους που έχουν ε, πολιτιστικά μνημεία κλπ. Επίσης, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη που απορρέουν για την ε, κοινότητα, για, την, ε, για τους πολίτες, για την οικονομία, μέσω της καλής διαχείρισης των, φυσικών, ε, των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Και του τουλεχθέντος είδαμε ότι υπάρχουν και σημαντικές απειλές σε αυτούς τους κοινού ε, χώρους, οι χώροι της φυσικής προστασίας αλλά και της πολιτικής κληρονομιάς αντιμετωπίζουν συχνά τα ίδια προβλήματα. Και γι' αυτό καταλήγουμε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και διαχείρισης αυτών των περιοχών. Και μιλούμε για περιοχές όπου όντως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τέτοιου είδου συνέργειε προ το κοινό καλό, το καλό όλων και για τη φύση και για τον πολιτισμό και την πολιτιστική μα κληρονομιά. Εδώ α πούμε μπορούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία, την συνειδητοποίηση, την εμπλοκή συμμετοχή των πολιτών και των κοινοτήτων σε αυτά τα project. Επίση, σε κάποια προγράμματα διαχείριση ε, των περιοχών αυτών, συνέργειε στην χρήση των διαθέσιμων πόρων, οικονομικών πόρων που υπάρχουν και όλα αυτά βεβαίω με στόχο όχι μόνο να διατηρήσουμε ή να αποκαταστήσουμε τις περιοχές αυτές, αλλά να ενισχύσουμε και το δυναμικό τους ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μεγαλύτερα ωφέλη, ε, διαθέσεις εργασίας ας πούμε ή για βιώσιμες δραστηριότητες. Εδώ να τονίσω ότι οι συνέργειες αυτές με τις ε, προστατευόμενες περιοχές του Natura 2000 έχουν σημαντικά ωφέλη, διότι στην Ευρώπη έχουμε ένα σημαντικό νομικό πλαίσιο το οποίο ακριβώς, στο οποίο ακριβώς βασίζονται αυτές οι, ε, αυτοί οι όροι προστασίας των ε, χωρών της, των περιοχών Natura 2000. Για το σκοπό αυτό, πέρσι υπήρξε ένα σχέδιο δράσης της Κομισιόν για την βελτίωση της εφαρμογής της, διατήρησης, ε, της, της νομοθεσίας για τη διατήρηση της φύσεως και έχουμε τονίσει την ανάγκη να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των, ε, του φυσικού και του πολιτιστικού κεφαλαίου, τονίζοντα φυσικά και το ευρωπαϊκό έτο. Ε, αυτή λοιπόν είναι η, συμβολή τη πλευρά του περιβάλλοντο στο ευρωπαϊκό έτο πολιτιστική κληρονομιά για το 2018. Ξεκινήσαμε κάνοντας κάποιες ε, μελέτες για να δούμε ποια είναι τα παραδείγματα που έχουμε όπου υπάρχουν τέτοιου είδους συνέργειες. Υπάρχει μια δημοσίευση με τις διάφορες ε, περιπτώσεις που μελετήσαμε από όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη και όντως είδαμε ότι υπάρχουν αρκετά, αρκετές συνέργειες, αρκετές δυνατότητες συμμετοχής και επικάλυψης. Ας πούμε, στη Ματέρα, στην Ιταλία, που θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της επόμενη, την επόμενη χρονιά. Υπάρχει, ε, αυτή είναι η περιοχή που είναι τμήμα της, ε, του δικτύου Natura 2000 και Βεβαίω ε, είναι πολύ γνωστή ω σημείο πολιτιστική, ω τόπο πολιτιστική κληρονομιά, ε, γιατί έχει πάρα πολύ σημαντικέ πολιτιστικέ αξίε και μνημεία. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι ωφελούν και τη διατήρηση της πόλης αυτής, αλλά και τα είδη πτηνών που χρησιμοποιούν ένα μέρος της ε, πόλης αυτής ως οικοσύστημα τώρα, τι γίνεται, τι βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν κάποιες μελέτε που γίνονται σε μεγαλύτερο βάθος. Προσπαθούμε να διαρευνήσουμε και, τα, και να κατανοήσουμε καλύτερα αυτέ τι χωροταξικές επικαλύψεις που υπάρχουν μεταξύ του, των ε, περιοχών Natura 2000 και των πολιτιστικών, της πολιτιστική κληρονομιάς Και προσπαθούμε μετά να αναλύσουμε και τις, ε, τους χώρους συνέργειας και να προτείνουμε καλές πρακτικές ε, για αυτή την ολοκληρωμένη διαχείριση, έχοντας βεβαίως πάντα υπόψη και τις ε, δυσκολίες, τις προκλήσεις σε ό,τι αφορά τον βιώσιμο τουρισμό, αλλά και τα ωφέλη που μπορεί να προκύψουν από όλη αυτή την προσπάθεια. Επίσης, Μέσω των αποτελεσμάτων που έχουμε από την έρευνά μας έχουμε καταγράψει ότι υπάρχει σημαντική επικάλυψη σε τόπους πολιτικής κληρονομιάς και Natura 2000 περίπου μισές από τις περιοχές πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται εντός ε, περιοχών Natura 2000 ή πολύ κοντά σε τέτοιου είδους περιοχές. Ας πούμε, από τις 336 ε, περιοχές ε, μοναδικές περιοχές ε, πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα μεγά, ένας μεγάλος αριθμός είτε επικαλύπτονται 100% ε, είτε βρίσκονται εντός 2 χιλιόμετρων από τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Κάτι παρόμοιο βλέπουμε εδώ, ακόμη πιο έντονο βέβαια, προκύπτει αν δούμε από τις, τις παγκόσμιες, τα παγκόσμια μέρη πολιτικής κοινωνίας από την UNESCO. Ε, σχεδόν όλα βρίσκονται σε περιοχές ε, μερικός ή ολικός ε, Natura 2000. Υπάρχει λοιπόν αυτή η επικάλυψη, η χώρο ταξική, την οποία είδαμε από τις πρώτες αυτές αναλύσεις που κάναμε. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες περιοχές επικάλυψης, ας πούμε, αυτοί που, αυτές που ε, ωφελούνται από ε, βραβεία από την ε, Europa Nostra. Πάλι οι μισές περιοχές που έχουν βραβευθεί από την Europa Nostra πάλι βρίσκονται εντός περιοχών Natura 2000. Αυτός λοιπόν είναι ένας τομέας όπου προσπαθούμε να προωθήσουμε τέτοιου είδου συνέργειες μέσω βραβείων που δίνονται για, ε, για την αριστεία στην διαχείριση από την Natura 2000 ή όταν εορτάζουμε την ημέρα Natura 2000 κάθε χρόνο την 21η Μαΐου. Επίσης ε, μίλησα και για κάποιους κοινού κινδύνους, κοινέ απειλέ που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές. Έχουμε διάφορα παραδείγματα πάλι καταγράψει. Οι απειλές αυτές είδαμε ότι είναι κοινέ. Ας πούμε, η μη βιώσιμη ε, διαχείριση από πλευρά τουρισμού ε, ή η ε, ανάπτυξη των πόλεων και η διαχείριση των υποδομών που γίνεται χωρίς σωστό σχεδιασμό. Αυτές λοιπόν οι απειλές μας δείχνουν και τις κοινέ προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτές τις περιοχές. Και ταυτόχρονα θέλουμε να τονίσουμε και τις ευκαιρίες που προκύπτουν όταν υπάρχει καλή, στοχευμένη, κοινή διαχείριση αυτών των περιοχών. Βλέπετε εδώ ένα ε, παράδειγμα από την Αυστρία. Υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης που λαμβάνει η υπόψη με σωστό τρόπο και την πολιτιστική αξία και την ανάγκη διατήρησης της, φυσικής, της φύσεως στην περιοχή εκεί. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στη φάση αυτή όπου προσπαθούμε να αναλύσουμε καλύτερα όλες αυτές τις προκλήσεις, τις απειλές και τις ευκαιρίες, έτσι ώστε να έχουμε συστάσεις και παραδείγματα καλών πρακτικών για να μας διευκολύνουν στην ε, καλύτερη πρόταση των ε, συστημάτων κοινή διαχείρισης. Και βεβαίως προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχουν ευκαιρίες για δημιουργία θέσεων εργασίας ή καλύτερη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής ή βιώσιμο τουρισμό, όπως τονίστηκε ότι είναι και ε, προτεραιότητα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έτους. Αυτές οι συστάσεις, τις οποίες εκπονούμε τώρα, θα έχουν ε, σχέση με την ε, καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα, με την καλύτερη επικοινωνία, με την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων, με την εξέβρεση μιας κοινή γλώσσας, συνεννόησης μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, γιατί νομίζω ότι προς το παρόν ε, μιλούμε λίγο παράλληλα οι διάφορες κοινότητες. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μια κοινή κατανόηση, ένα κοινό σκεπτικό, και βεβαίω να υπάρχει καλύτερη ε, ενσωμάτωση όλων αυτών των στοιχείων στην πολιτική, να υπάρξουν κοινέ πρωτοβουλίε και καλύτερη ευαισθητοποίηση των κοινωνικών οικονομικων ωφελών που μπορούν να προκύψουν από αυτές τις κοινέ ε, δυνατότητε διαχείρισης αυτών των περιοχών. Και επίσης καλύτερο σχεδιασμό και σε άλλου τομεί που μπορεί να επηρεάσουν αυτές ε, τις κοινέ περιοχές. Μίλησα για τον τουρισμό, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς που επηρεάζουν, α πούμε, ε, η ανάπτυξη τη υπαίθρου. Και επίση, όλες αυτές τις καλέ πρακτικές θέλουμε να μπορούμε να τις ανταλλάξουμε στις, μεταξύ, να τους ανταλλάξουν οι διάφορε κοινότητε μεταξύ τους και θέλουμε να καταγράψουμε την ανάγκη που υπάρχει για αλλά και τι διαθέσιμε ευκαιρίες χρηματοδότησης κυρίως μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων έτσι ώστε να μπορούμε αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι έχει λοιπόν η κατάσταση. Υπάρχει και ένα φυλάδιο το οποίο μπορείτε να πάρετε αν θέλετε να δείτε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής γιατί θεωρούμε ότι το μέσο αυτός μας δίνει πολύ σημαντικές ευκαιρίες για τη δημιουργία συνεργειών και για αμοιβαία ωφέλη για την κοινή μας δουλειά. Σας ευχαριστώ. Merci. Acum ultimul ε, intervenient, domnul Oriol Matalonga de la UNESCO. Ο κύριος Οριόλ Ματαλόγκα από την UNESCO, τελευταίος αγορητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διάκονο για την πρόσκληση. Ας πάμε σε μια άλλη γλώσσα του Νότου, την Ισπανική. Να σας μιλήσω λοιπόν στα Ισπανικά ως ε, αντικατοπτρισμό της ε, γλωσσικής και πολιτικής πυκλομορφίας Ευρώπης. Βέβαια εγώ την παρουσίασή μου την έχω, κάνει, την έχω ετοιμάσει στα αγγλικά οπότε θα αρκετά μίλησα. Θα μιλήσω κάποια στιγμή και αγγλικά μάλλον. Είναι μεγάλη χαρά για την UNESCO να βρισκόμαστε εδώ μαζί σας σήμερα. Εκπροσωπώ μια οργάνωση που έχει στην καρδιά της ε, την πολιτική κληρονομιά, μάχεται για αυτήν. Αυτή τη μοναδική στιγμή είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτό το κοινό μας έργο υπέρ της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς. Ε, ιδιαίτερα δε κατά τη διάρκεια αυτού του εξαιρετικού έτους ευρωπαϊκής πολιτικής κληρονομιάς. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια πράγματα, κάποια προγράμματα τα οποία έχουμε σε πόλεις και σε περιοχές στις οποίες η UNESCO συνεργάζεται με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του ε, τους που γιορτάζουμε την πολιτική κληρονομιά. Και τώρα από εδώ και πέρα να μιλήσω λίγο στα αγγλικά γιατί έχω ετοιμάσει τα αγγλικά την παρουσίασή μου. Για τη συνεργασία μεταξύ UNESCO και Ευρωπαϊκής Ένωσης νύχτα, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Όπως γνωρίζετε η UNESCO έχει μια μακρόχρονη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ε, πολιτισμού, ε, παιδείας ε, και έρευνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στρατηγικό σύμμαχος της UNESCO, είναι δύο οργανώσει που μοιράζονται τι ίδιε αξίες και συνεργάζονται στενά για να πετύχουν κοινού στόχους. Σε ό,τι αφορά το θέμα που συζητούμε σήμερα, την πολιτική κληρονομιά, πάνω από 350 σημεία πολιτική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και σημεία πολιτικής, πολιτική κληρονομιά τη της UNESCO. και πολλά από αυτά επίσης είναι ε, εγγεγραμμένα και στον κατάλογο της άειλης πολιτικής χρονιάς UNESCO. Η Το Ευρωπαϊκό Έτος λοιπόν είναι μια ευκορία, ε, ευκαιρία για να καταγράψουμε την πολιτική κληρονομιά ως ακρογωνία ολίθο του ευρωπαϊκού οράματος, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του μέλλοντος να θυμάστε ότι η δημιουργικότητα και η πολιτική κληρονομιά είναι αλληλένδετα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και ο πολιτισμός είναι ο στόχος μας. Η UNESCO με χαρά έχει συνεργαστεί στενά με όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, σε, όλα αυτά τα, σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που ανέφερε η Ερμήνια αλλά και με άλλες γενικές διευθύνσεις όπως η, Γενική Διεύθυνση Grow αλλά και στη διεθνή διάσταση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτική Ονομιάς, η καταπολέμηση του παρανομού εμπορίου Έχουμε μια σημαντική πρωτοβουλία για την εφαρμογή του νόμου. Συναντιόμαστε στο Παρίσι με, τους, με, εισαγγελείς ε, και τελωνιακούς για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα. Το θέμα της παράνομης διακίνησης και εμπορίας πολιτικών αγαθών είναι τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για όλη την ευρύτερη περιοχή και όλο τον κόσμο γενικότερα. Αυτά για τη διεθνή σχέση, ε, διάσταση. Ε, Επίση ασχολούμαστε σε, με θέματα πολιτική οικονομία σε κίνδυνο με την Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση την Γεμένη, την Σύρια, τη Λιβύα, το Ιράκ, την Κεντρική Ασία. Είναι τεράστιος ο αριθμό των προγραμμάτων στα οποία συνεργαζόμαστε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο τη Ευρώπη συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΟΚΕ, η Επιτροπή των Περιφερειών, είναι όργανα με τα οποία συνεργαζόμαστε. η Αρμίνια το είπε και προηγουμένως ότι 19 όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρμοδιότητες ε, για το θέμα της πολιτικής χρονομιάς αλλά και διαθεσμικά, διοργανικά, όπου όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται μεταξύ τους και με την UNESCO, ε, είναι ο τρόπος εργασία προκειμένου να εξασφαλίσουμε αυτή τη σφαιρική προσέγγιση. Ο κ. Διακονού και ε, τα μέλη της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Παιδείας ιδιαίτερα Μα έχουν ιδιαίτερα βοηθήσει γιατί έχουν στηρίξει την UNESCO. Αυτή η πρωτοβουλία για την οποία θα σα μιλήσω ε, έγινε κατορθωτή χάρη σε μια δράση προετοιμασία τη επιτροπή αυτή που υλοποιήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Growth τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχο είναι να προωθηθεί και να αξιοποιηθεί η πολιτική κοινωνία στην Ευρώπη μέσω του πολιτικού τουρισμού και μέσω μια συμμετοχική και σφαιρική προσέγγιση. Τι σημαίνει αυτό. Βλέπετε είναι η Γκάρ, η γέφυρα της Γκάρ στη Γαλλία. Είναι παγκόσμια πολιτική κληρονομιά. Σύντομα θα έχετε αυτή τη φωτογραφία να μπορείτε να την κατεβάσετε στα κινητά σας τηλέφωνα, ε, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη ένα link σε αυτό το site, πολύ χρήσιμο, ε, τι είναι τα ταξίδια παγκόσμια κληρονομιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο τίτλο ε, του, του προγράμματο αυτού. Είναι μια πλατφόρμα η οποία αναπτύσσεται σε συνεργασία με, το, με την National Geographic που παρουσιάζει ένα καινούριο τρόπο να ε, ταξιδέψει κανείς σε όλα τα ε, σημεία πολιτική, παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας στόχος είναι ε, αγαθά πολιτικής, παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι πολύ γνωστά αυτή τη στιγμή, να γίνουν πιο γνωστά, να προβληθούν και ε, να γίνουν πιο γνωστά. Για να εμπνεύσουμε λοιπόν τους ο, ταξιδιώτες ε, ε, υιοθετήσαμε τέσσερα τέσσερις πυλώνες, τέσσερις άξονες. αρχαία Ευρώπη, Ρωμαντική Ευρώπη, Βασιλική Ευρώπη και υπόγεια Ευρώπη. Μέσω αυτών των ταξιδιωτικών διαδρομών θα ανακαλύψετε την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα καινούριο, υπό ένα καινούριο φως, ε, υπό ένα καινούριο πρίσμα και κάθε μία αυτές τις διαδρομές θα διηγείται διαφορετικές ιστορίες προσπαθούμε να προβάλλουμε τους, ε, τα, χαμένα, τα, τα κρυφά διαμάντια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Χρονομιάς και συνεργαζόμαστε με τις τοπικές επιχειρήσεις, με τους ενδιαφέρομενους φορείς, με τις αρχ, τοπικές αρχές. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ταξιδεύουν στον, ε, στην, ε, στα πολιτικά αγαθά. Να επιμικηθεί η ε, διαμονή τους, ε, να, οι τουρίστες να επισκέπτονται περισσότερες περιοχές κλπ. Αυτό το πρόγραμμα ε, αναπτύχθηκε με 34 σημεία πολιτικής χρονιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε έρθει σε επαφή με, με τις τοπικές αρχές, τους, τοπικούς επιχειρηματίες κλπ. Αρχές ε, διαχείρισης, ε, επιμελητήρια, τουριστικά επιμελητήρια, τους εκπροσώπους ε, των ξενοδοχειακών μονάδων, τις τοπικές κοινότητες, τους εμπειρογνώμονες τουριστικής βιωσιμότητας. Όλοι αυτοί έχουν συνεισφέρει με έναν τρόπο πάρα πολύ χρήσιμο. Ε, η υψηλό επίπεδο διάσκεψη για τον ε, βιώσιμο τουρισμό που έλαβε χώρα πριν από δύο εβδομάδε στο Παρίσι ε, στα, στο αρχηγείο της UNESCO σχετίστηκε με αυτό ακριβώς το θέμα και με το έτος τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας που είναι το 2018 εντοπίστηκαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο βιώσιμος πολιτικός τουρισμός και το λύσεις για το πώς θα ξεπεραστούν. Αυτό το πρόγραμμα ε, είναι το πρώτο το οποίο σχετίζεται με τον βιώσιμο πολιτικό τουρισμό ε, από το Σεπτέμβριο 2018 βγήκε στο ίντερνετ, ξεκίνησαν εκστρατείε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 34 ε, σημεία παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς στην Ευρώπη λοιπόν συμμετέχουν σε τέσσερις άξονες ε, θα ήταν μόλις, μόλις ολοκληρωθεί θα σα το, θα σας κάνουμε μια επίδειξη θα ήταν πολύ καλό τώρα δύο λόγια για τη σύνδεση αυτή μεταξύ πολιτικής κληρονομιάς και τουρισμού. Ο τουρισμός είναι ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους της ε, παγκόσμιας οικονομίας. Έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει άμεσα ή έμεσα σε πολλούς από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Μην ξεχνάτε την Ατζέντα 2030 είναι πολύ σημαντική σε καθημερινό επίπεδο. Ο πολιτικός τουρισμό αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή το 40 σχεδόν της των εισοδημάτων από τον τουρισμό συνολικά. Και το 10% του συνολικού παγκόσμιου πλούτου. Αν το διαχειριστούμε αυτό τον τουρισμό υπεύθυνα και βιώσιμα, μπορεί να προστατεύσει την πολιτική κληρονομιά και να προωθήσει την δημιουργικότητα σε όλες τις μορφές. Ε, τα, ε, ε, οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν παν, ε, σημεία παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς ε, χαρακτηρίζονται από δημιουργία πολλών θέσεων απασχόλησης επίσης. το, τα ταξίδια αυτά είναι ταξίδια ε, δύο χιλιετιών και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και ιδίω νέοι που θα θέλανε να τα διατρέξουν όλα. Με αυτή την εφαρμογή αυτό θα γίνει δυνατό. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ, Λίγο Πρόεδρος. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις και μία από αυτές θα μπορούσε να είναι ότι Ίσως αυτό που έχουμε προβλέψει στο πρόγραμμά μας ε, ε, ερωταπαντήσεις να μην είναι επαρκές, γιατί δεν είναι πλέον καν θέμα απλώς ερωτήσεων. Ε, ε, πρόκειται για απόψεις, για οπτικές γωνίες, για ενημέρωση που αφορά στην πραγματικότητα που, που είναι πολύ διαφορετική μεταξύ των κρατών μελών, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε, να αναφερθούμε πολύ και στο θέμα της διαφορετικότητας. Δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε το επόμενο βήμα να προστατευτούμε δηλαδή την πολιτιστική μας κληρονομιά χωρίς να κατανοήσουμε καλύτερα τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αναλάβουμε δράση. Περιμένω λοιπόν όχι μόνο τις ερωτήσεις σας αλλά και τις απόψεις σας και την δική σας προσέγγιση. Μαρία Γκούστα Σάντους από το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας και μέλος της Επιτροπής ε, Παιδείας και Επιστήμης. Η Πορτογαλία συνεχώς ε, προσπαθεί να εστιάζεται στην προώθηση και σε μελέτες τεχνικές και επιστημονικές για θέματα πολιτικής χρονιάς σε συνεργασία με επιστημονικά έρευνα. Αυτό μας επιτρέπει να γνωρίζουμε καλύτερα και σε περισσότερο βάθος την πραγματικότητα της πολιτικής κληρονομιάς στην Πορτογαλία. Βασιζόμαστε σε τρεις ομάδες που είναι ειδικευμένε. Ε, το εργαστήριο συντήρησης Ζωζέντε Φεγγερέδου, το εργαστήριο τέχνης και το εργαστήριο ε, ε υποβρύχιας ε, αρχαιολογίας. Όλα αυτά ε, μας έχουν βοηθήσει να κάνουμε σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Του χρόνου θα κάνουμε Εθνικό Μουσείο Αντίστασης ε, το κάστρο της, το κρατηρίου Πενίσε. Είναι ένα από τα παραδείγματα για το μέλλον. Επίσης ε, κινητοποιούμε ευρωπαϊκά κονδύλια, απλοποιούμε τις ε, διαδικασίες για παρεμβάσεις ε, σε τοποθεσίες πολιτικής χρονομιάς κλπ. Χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση της πολιτικής μας χρονομιάς. Αυτό είναι σαφές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήταν ο τιμονιέρης αυτής της διαχείρισης τα τελευταία χρόνια. Ο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξάρτητα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια πρόκληση την οποία θα πρέπει, στην οποία θα πρέπει να απαντήσουμε όλοι μαζί. Σε αυτή την ε, πορεία, κοινή μας πορεία, θα πρέπει να εστιάσουμε στις ανάγκες των πολιτών και στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, αξιοποιώντας την αξίε του, της ευρωπαϊκής πολιτικής και με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές είναι οι προσδοκίες που έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μας βοηθήσει στη διαχείριση πολιτικής μας κληρονομιάς. Ευχαριστώ. Και πάλι καλό απόγευμα σε όλους. Ε, ε, λυπούμε που επανέρχομαι, αλλά υπάρχει μια σκέψη που δεν θα ήθελα να την έχω αφήσει χωρίς αναφορά στη σημερινή συζήτηση. Εμείς, εγώ λοιπόν προέρχομαι από μια μικρή περιοχή, η οποία όμως ε, είναι στην ε, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO εμπίπτει σε όλα τα χαρακτηριστικά και στοιχεία που αναφερθήκαμε για την φυσική και για την περιβαλλοντική δηλαδή και την πολιτισμική κληρονομιά. Πρέπει λοιπόν η εθνική, η ευρωπαϊκή και οι διεθνή φορείς να συνεργαστούν καλύτερα προκειμένου να προστατευτούμε την πληρονομία αυτή. Αλλά πολύ συχνά κάνουμε ένα λάθος ίσως λόγω μιας προσέγγισης των πολεοδόμων ή άλλων ρυθμιστών. Ε, δηλαδή τα, τα μεταχειριζόμαστε με, τρόπο τελείως απομονωμένο από το φυσικό και αστικό τους περιβάλλον και σαν να είναι ε, θησαυροί που δεν πρέπει να τους πολυακουμπάει κανείς εγώ πιστεύω ότι ο συσχετισμό των αγαθών αυτών της πολιτιστικής κληρονομιάς με τους κατοίκου τη περιοχή με τους επισκέπτε και κάτι που θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και που θα ήταν και πλεονέκτημα οικονομικό είναι η καλύτερη αρμονική σχέση των τεχνητών που θα χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των μνημείων, την ε, προστασία των, ε, των δομών που τα προστατεύουν κτλ. Και σε μια συνολική προσέγγιση που θα πρέπει να προσελκύει επισκέπτες. Δεν μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε τα μνημεία χωρίς να σκεπτόμαστε τον πληθυσμό, τους κατοίκους της περιοχής και τις οικονομικές τους ακόμα ανάγκες δεν θα μπορούσαμε να μιλούμε για Ευρω... Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχουμε μια συμβίωση που είχαμε όλους αυτούς τους αιώνες και που μας οδηγεί στην, στην ανάγκη της προστασίας τους και δικαίως αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ε, με ενδιαφέρει να συνεχίσω την ε, σκέψη του συναδέλφου. Ε, εγώ προέρχομαι από την ε, Ελλάδα οι, τα αστικά κέντρα έχουν κενά τα οποία τα δημιουργούν τα ευρήματα, τα αρχαιολογικά. Έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα και συγκροτήματα εκτός ε, πόλης, στην Ήπεθρο. Άρα σχετίζεται το κληροδότημα, το πολιτιστικό κληροδότημα, με τον πολεοδόμο, με τον χωροτάκτη, με τον αγρότη, με τον ε, ε, κλέφτη δηλαδή με αυτόν που θα εκμεταλλευτεί τις αφύλακτες αυτές ε, ενότητες ε, και θα μπορέσει να τις εμπορευτεί. Το ζήτημα της προστασίας για το οποίο συζητάμε και στο οποίο τοποθετήθηκα και προηγουμένως, επίσης έχω και ενάλλειες αρχαιότητες, ε, πάρα πολλά ναυάγια, και επομένως το ζήτημα της ασφάλειας, της εποπτείας είναι κρίσιμο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε μόνο να επενδύουμε μόνο στην ανταλλακτική σημασία και μόνο στην ανταλλακτική και οικονομική σημασία ή σε μια μεταφυσική που θέλει να μας κάνει να συσχετιστούμε με το παρελθόν μας και να νιώθουμε υπερήφανοι γι' αυτό. Πρέπει να βρούμε νέα μεικτά πρωτόκολλα. Το νέο δίκαιο που χρειάζεται να συσταθεί και το οποίο πρέπει να είναι ευλίγιστο και η ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τα εργαλεία να το εισηγηθεί. Το νέο δίκαιο πρέπει να είναι να βοηθάει και τη συσχέτιση του ευρήματος με τον πολίτη, αυτό που είπε ο συνάδελφος, με την καθημερινή του ανάγκη, με την καθημερινή του πράξη και επίσης να, προτείνει τρόπους νομιμοποίησης του ιστορικού ευρήματος, του πολιτιστικού ευρήματος. Η βαθύτερη προστασία δεν είναι πια μόνο ε, χημική. Η βαθύτερη προστασία είναι πολιτισμική είναι να μπορέσουμε να δεχτούμε το κληροδότημα ως οργανικό κομμάτι της ζωής μας και όχι ως ένα απόμακρο και αποσπασμένο κομμάτι που αντιστοιχεί στην ιστορία και που κάποιοι τουρίστες μπορούν να το ε, επισκεφτούν. Αυτή, αυτό νομίζω είναι το κλειδί και με συγχωρείτε αν ε, μακρηγορώ αυτό νομίζω είναι το κλειδί στο οποίο πολιτικά ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εισηγηθεί λύσεις. În mod excepțional, acest subiect Κατά εξαίρεση, η δικτατορία δεν ε, δουλεύει. Έχουμε τελικός χρόνο, αλλά αυτά που είπατε στις παρεμβάσεις σας θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν και νομικοί και συνέπειες. Ε, ίσως όντως να χρειάζεται και μια νομική εδώ παρέμβαση. Ο κύριος Μεντόλα μάλλον είναι ο καθήλυν αρμόδιος, είναι εδώ από την νομική υπηρεσία του, του Κοινοβουλίου, οπότε μπορείτε να πάρετε το λόγο και να μας διαφωτίσετε. Yes, thank you. Good evening. Ε, Giovanni Mendola. Ε, Giovanni Mendola από την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως υπόθηκε πολλές φορές σήμερα, η πολιτική κληρονομιά και η διατήρησή της είναι όντως ένα θέμα με το οποίο ασχολούνται αποκλειστικά τα κρατημέλη. Αλλά υπάρχουν και κάποιες πτυχές οι οποίες αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω ότι στα πλαίσια του άρθρου 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ένωση θα εξασφαλίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά διασφαλίζεται. Και στο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγεται ότι την αρμοδιότητα ώστε η πολιτιστική κληρονομιά να προωθηθεί έχει δοθεί, την, έχουμε, την έχει αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση που διασφαλίζει την πολιτιστική κληρονομιά. Ο κανόνας αυτός εισήχθη από την συνθήκη του Μάστριχτ, αλλά ακόμα και πριν το Μάστριχτ η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα δρούσε στα πλαίσια της ε, διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως γενική αρχή. Αναφέρθηκαν διάφορες αρχές πιο πριν ε, για, την, ε, ε, το εμπόριο των πολιτιστικών αγαθών που ήταν κομμάτι αυτών των πρωτοβουλειών πριν το Μάστριχτ, παρόλο που μπορεί να βασίζονται σε διαφορετικές νομικές βάσεις, όπως κυρίως η εμπορική πολιτική. Η διατήρηση λοιπόν της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι συναρμοδιότητα. Υπάρχει λοιπόν η αποκλειστική αρμοδιότητα και η συναρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό. Και βεβαίως αυτή είναι η λιγότερο ισχυρή, αν μπορώ να το πω έτσι. Η αρμοδιότητα αυτή έχει να κάνει με την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αλλά και με την στήριξη και τη συμπλήρωση των δράσεων των κρατών μελών. Πέραν λοιπόν το ότι είναι συμπληρωματική αρμοδιότητα, το δικαστήριο από την αρχή, και εδώ πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο ο που είναι συμπληρωματική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η εκπαίδευση και ο αθλητισμός. Επίσης, η προστασία της υγείας, η πολιτική προστασία, η διοικητική συνεργασία, η βιομηχανία και αυτοί οι τομείς αποτελούν συμπληρωματικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαστήριο λοιπόν πάντα υπογράμμιζε ότι το γεγονός ότι μία αρμοδιότητα έχει συμπληρωματική φύση δεν σημαίνει ότι δεν είναι αρμοδιότητα. Υπάρχει αρμοδιότητα και εφόσον υπάρχει αυτή η αρμοδιότητα, παρόλο που είναι συμπληρωματικής φύσεως, οι γενικές αρχές εξακολουθούν να ισχύουν. Οι οριζόντιες αρχές λοιπόν στον ε, τομέα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ο κανόνας επίσης της ειλικρινού συνεργασίας των κρατών μελών ισχύει που σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, απόσχουν από υιοθέτηση μέτρων που μπορεί να ε, δυσκολέψουν την επίτευξη των στόχων που θέλει να επιτύχει η ευρωπαϊκή πολιτική. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασκεί τις αρμοδιότητές της. Παρόλο λοιπόν που δεν υπάρχει άμεση ρυθμιστική ισχύ σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση αρμοδιοτήτων, όπως υπάρχει σε άλλους τομείς, εσωτερική αγορά για παράδειγμα, η ενωσιακή αρμοδιότητα υπάρχει, υφίσταται και μπορεί να ασκηθεί κυρίως για να στηρίξει τις δράσεις των κρατών μελών. Επίσης, κάτι άλλο θετικό είναι ότι υπάρχει μια πολύ θετική στάση του συστήματος απέναντι στην χρηματοδότηση πρωτοβουλειών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περιλαμβανομένου και ενός τομέα που είναι πραγματικά πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το δίκαιο του ανταγωνισμού στα πλαίσια του 107 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αδειοδοτήσει την κρατική ενίσχυση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ακόμη και όταν διακυβεύονται οικονομικές δραστηριότητες. Ε, για να μην μιλήσουμε για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα ή διάφορα τέτοιου είδους project σε αυτή την περίπτωση εκπίπτουν αυτά του, παιδι, του πλαισίου της ε, κρατικής επιχορήγηση. Οπότε η κρατική αυτή ενίσχυση για την στήριξη της πολιτιστική κληρονομιάς καλύπτεται και από τον, κανονισμό, τον γενικό κανονισμό για τις συνολικέ εξαιρεσει. Στον τομέα λοιπόν αυτό, ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, συμπληρωματική αρμοδιότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα. Και εφόσον τα κρατημέλη είναι διατεθειμένα να ολοκληρώσουν τέτοιου είδους δράσεις που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί έχουν μεγάλο περιθώριο ελιγμών σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κατ' της Α, ή μάλλον ο κύριο Μέντολα όταν θέλει να ξαναπαρέμβει μπορεί να μου το πει. Σα ευχαριστώ Ραφέλ Ζεγά από το Γαλλικό Κοινοβούλιο για τα θέματα πολιτισμού και παιδεία. Εμείς έχουμε μια παλαιότατη πολιτική και νομίζω ότι είμαστε μεταξύ των χωρών εκείνων που έχουν τα νομοθετικά εργαλεία τα πολύ στοχευμένα στη διάθεσή τους για τα θέματα της προστασίας πολιτισμού αλλά και το δικό μας ε, σύστημα βασίζεται ε, στην ε, εγγραφή στα μητρώα των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό συνδέεται με αυτό που έλεγε και ο αυστριακός συνάδελφος νωρίτερα. Και προετοιμάζουμε και μία μελέτη για τα έργα αποκατάστασης ε, των ήμιων αυτών και δεν μιλούμε μόνο για τα αναγνωρισμένη ε, αρχιεκτονικής και ιστορικής σημασίας νημεία, αλλά την προστασία ε, της ταυτότητάς τους αλλά και την ε, περιοχή στην οποία βρίσκονται, ε, της πόλεως ή της υπαίθρου. Τώρα ανεφερθήκατε και στις έντονες πιέσεις που ασκούνται από οικονομικά συμφέροντα ή πολιτικά συμφέροντα που δεν έχουν αναγκαστικά την ίδια ανησυχία ή το ίδιο ενδιαφέρον για τα μνημεία του πολιτισμού που έχουμε εμείς εδώ και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι πρέπει να επαγρυπνούμε διαρκώς στην εφαρμοσιμότητα και την ε, ευελιξία των διατάξεων αυτών που πρέπει να έχουν δηλαδή γιατί έχει δείξει η υλοποίηση της πολιτικής μας και τα όρια της ε, και πολύ συχνά βρισκόμαστε σε μια συνολικά καλή κατάσταση ε, προστασίας των μνημείων, φυσικής προστασίας αλλά πολύ συχνά δεν έχουμε ε, επαρκείς λύσεις ε, επανάχρησης ε, αποκαταστημένων κτίριων. Γνωρίζουμε ότι ένα ιστορικό κτίριο, ένα ιστορικό μνημείο που δεν συντηρείται επαρκώς μετά από 15-20 χρόνια απαιτεί νέα αποκατάσταση. Στη Γαλλία λοιπόν εξετάζουμε αυτή τη στιγμή τα προβλήματα αυτά μέσω μιας προσέγγισης ε, που την ονομάζουμε σχέδιο δράσης ε, για τα κέντρα της πόλεως σχετικά με περιοχές που έχουν ε, απολέσει αν θέλετε το κοινωνικό και οικονομικό τους ακόμη ενδιαφέρον μέσα στο πλαίσιο του αστικού ιστού επανεισαγάγοντας βεβαίως και τη σημασία, όπως λέγατε και εσείς ε, ε, Πρόεδρε και ε, οι υπόλοιποι ομιλητές, η κυρία της Κομισιόν, για τους τεχνίτες που ασχολούνται με την αποκατάσταση, για άλλους τεχνίτες που ασχολούνται με την οικοδόμηση και μάλιστα την λεπτή οικοδόμηση που απαιτούν αυτά τα μνημεία, που τους απαιτούμε απολύτως, τους χρειαζόμαστε απολύτως και ώστε να του συνδυάζουμε με την υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα που θα περιβάλλει αυτά τα μνημεία. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω ποιο άλλο θα ήθελε το λόγο, παρακαλώ. Okay. Um, so good afternoon. name uh, ε, καλό απόγευμα σε όλους από το Μαριστήμιο του Λόβεν είμαι και μέλος ε, του Συμβουλίου Ευρώπα Νόστρα και είμαι υπεύθυνο ενό ε, από το πάνελ ε, που απονέμει βρα, βραβεία που, στα οποία αναφερθεί και νωρίτερα σε πόλεις μεγαλύτερες και μικρότερες. Μπορώ να σας πω ότι εμείς καταγράφουμε μία τάση όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι είναι όλο και πιο σημαντικοί στην προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί πολύ συχνά δίνουμε το βάρος της προσοχής μας στα ίδια τα συγκροτήματα, τα κτηριακά, τα μνημεία, αλλά πρέπει να προσέχουμε όλο και περισσότερο τη διασύνδεση με την τοπική κοινωνία. Εμείς λοιπόν ε, έχουμε και την Προεδρία της UNESCO στην ε, προληπτική αποκατάσταση όπως την ονομάζουμε ε, γιατί αυτό στο οποίο στοχεύουμε είναι να έχουμε ένα ε, σύστημα υγείας αν θέλετε των μνημείων αυτών που δεν είναι σαν την προληπτική υγεία είναι μια πιο συστηματική προσέγγιση που θα μας επέτρεπε να διανεργούμε και έρευνες και μελέτες εκ μέρους και, και λογαριασμό δημόσιων φορέων όπως το Συμβουλίο της Ευρώπης αλλά δεν είναι στόχος καθεαυτός και από μόνος του χρειάζονται συνδυασμοί διαφόρων πόρεων και διαφόρων προσεγγίσεων και νομίζω ότι αυτό που ήδη ελέγχθη σήμερα αρκετέ φορές είναι πώς προσμετρά κανείς, πώς αξιολογεί τις επιλογές που πρέπει να κάνει, που καλείται να κάνει. Και ένα πρόβλημα που συχνά αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ευρώπη είναι ότι προσμετρούμε, μετράμε μόνο οικονομικά. Μόνο χρηματοοικονομικά. Δεν μετράμε την αξία του περιβάλλοντος ή την κοινωνική αξία ή άλλες διαστάσεις που μπορεί να έχει ως σημασία ε, οποιοδήποτε τόπος, το οποιοδήποτε μνημείο, προκειμένου να αξιολογήσει κανείς, να εκτιμήσει πληρέστερα τη σωστή θέση που θα πρέπει να κατέχει και τους σωστούς πόρους που θα πρέπει να αποδίδονται ή στην πολιτιστική κληρονομιά. Ε, πολλά μπορεί να προσθέσει κανείς, αλλά ε, ένα από τα στοιχεία που και την περασμένη εβδομάδα που ήμασταν στην συνάντηση και συζητούσαμε ε, ε, και θα έπρεπε ίσως να αναφέρουμε περισσότερο, είναι πράγματι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι, οι πολίτες. Αναφερόμαστε στις δεξιότητες, αλλά οι δεξιότητες είναι άχρηστες αν οι γονείς που μεγαλώνουν τα παιδιά δεν πείθονται ότι πρέπει να οδηγήσουν το παιδί τους προς την συγκεκριμένη ας πούμε ειδίκευση. Δηλαδή αν ε, σταματήσουν οι γονείς να θεωρούν ότι τα παιδιά τους πρέπει να γίνονται γιατροί, θα γίνονται υδραυλικοί. Για να πω ένα απλοϊκό παράδειγμα. Δηλαδή, ε, η ευαισθητοποίηση περνάει από πάρα πολλά επίπεδα σχετικά με το πόσο μπορεί να καλύπτει ένας άνθρωπος τη φιλοδοξία του διοχετευόμενος προς συγκεκριμένη ειδικότητα επαγγελματική. Και αυτό πρέπει να το προσέχουμε επίσης. Και κοιτώντα του διάφορου χρηματοδοτικού μηχανισμού που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσω να ήταν πολύ καλή ιδέα να λάβουμε υπόψη μας ε, σχετικά με τα θέματα της προστασίας της ταυτότητας και του πολιτισμού της Ευρώπης ε, είναι η αντίληψη αυτών των ε, ενιών εις τους πολίτες, στην κοινή γνώμη, στην πλειοψηφία των πολιτών. Ο καταλληλότερος τρόπος λοιπόν προστασίας των μνημείων είναι η όλο και πιο προσεκτική επένδυση στις κοινωνίες. Τα καλύτερα παραδείγματα που έχουμε για την προστασία και καλή λειτουργία ιστορικών μνημείων είναι αυτά που περιβάλλονται από μια ενεργητική τοπική κοινότητα που λειτουργεί και σε οικονομικό επίπεδο πλήρως και επαρκώς. Και αυτό ε, κάνει υπό μια έννοια κανείς και μέσω του Natura 2000 θα μπορούσαμε να δούμε την Natura 2000 για το πόσο είναι σημαντική για την υγεία μας την ίδια και για το πόσο προστατεύει ή υποστηρίζει την μετανάστευση των πτηνών αλλά όχι, γιατί όχι και των ανθρώπων με τις δεξιότητες τους, με τις επαγγελματικές τους προτιμήσεις κτλ. Αυτό θα, θα συνεισέφερε προς την προστασία της ταυτότητας ε, της Ευρωπαϊκής. Και για τα European Heritage Awards ε, νομίζω ότι θα βλέπαμε πολύ χρήσιμα, πολύτιμα παραδείγματα που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε ως Ευρώπη. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Ε, ε, θα ήταν καλό να γίνει μια... να εξετάσουμε μάλλον ε, την περίπτωση να κάνουμε μια καινούργια μελέτη. Ε, μάλλον πριν από δύο χρόνια μιλούσαμε ήδη εμείς για την σφαιρική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς σε μια έκθεσή μας. Θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά ξανά σε αυτή την έκθεση που είχαμε κάνει πριν από δύο χρόνια. Ε, και νομίζω ότι ήδη από τότε μιλούσαμε για τη σημασία της διαχείρισης πολιτικής κληρονομιάς προς όφελος του τοπικού πληθυσμού. Παρακαλώ, κυρία μου, εσείς. Θέλετε το λόγο. Σηκώσατε το χέρι σας. Παρακαλώ. Uh, Προέρχομαι από το Κοινοβούλιο της Σερβικής Δημοκρατίας. Ε, θα ήθελα να ε, συγχαρώ όλους τους συναδέλφους που μίλησαν Παρακολούθησα με προσοχή τα όσα υπόθηκαν και τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Για όλους μας η προστασία της πολιτικής χρονιάς είναι πρώτη προτεραιότητα. Πριν από μερικές μέρες στη Σερβία οθετήσαμε ένα καινούριο νόμο για την προστασία των μνημείων μας. Ε, ο πόλεμος πια είναι στο παρελθόν της ιστορίας μας. Παρόλα αυτά άφησε πολλές πληγές. Και διδαχθήκαμε πολλά πράγματα. Θέλω να επιστήσω τους προσοχή σας σε ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε στο, στο Νότο, στο Μετόχι και στο Κωσυφοπέδιο πεδίο βλέπουμε συστηματική καταστροφή χριστιανικών μοναστηριών, εκροταφείων και εκκλησιών. Και θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. 14 χρόνια μετά την καταστροφή 25 ε, περίπου εκκλησιών, χριστιανικών εκκλησιών ε, το 2004. Είναι δυνατόν στην Ευρώπη να δεχόμαστε χωρίς καμία απάντηση την καταστροφή αυτής της πολιτικής χρονομιάς, χωρίς κανείς να ξέρει την ταυτότητα των υπετίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής ε, ε, Πολιτισμού στην Βουλή της ε, Βιέννης και είμαι και ιστορικός. Και συνήθως ως ιστορικός με ανοιχτά μάτια κοιτώ την πόλη μου και τίθεται το ερώτημα ποιος προσέχει την πολιτιστική κληρονομιά, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το θέμα. Στην Αυστρία υπάρχει μια ιεραρχία. Έχουμε ένα Ινστιτούτο το, της, ε, το Ομοσπονδιακό, το οποίο όμως ε, ασχολείται και προστατεύει χιλιάδες ε, μνημεία. Και βεβαίως έχει πάρα πολλή δουλειά και υποχρεώσεις. Επίσης, οι ιδιοκτήτες ίσως θα καλό θα ήταν να προσέχουν τα πολιτιστικά τους μνημεία ή κτίρια. Οπότε το θέμα είναι πάντα ποιος προσέχει αυτά τα μνημεία. Και θα ήθελα και την άποψη των νομικών. Γιατί εκεί, όπως είπε ο εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας, υπάρχει συμπληρωματική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως λοιπόν αυτό εδώ να είναι σημαντικό για το ποιος δηλαδή παρεμβαίνει και ποιος φροντίζει την πολιτιστική κληρονομιά ενσυνείδητα. Γιατί το ε, Ομοσπονδιακό Γραφείο των α, Πολιτιστικών Μνημείων πραγματικά έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, έχει πάρα πολλά μνημεία να προστατέψει, να προσέξει και πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους βοήθεια. Μπορώ να θυμηθώ, τώρα που μίλησε η ε, συνάδελφος από τη Σερβία, ότι τελευταία 40 χρόνια έχουν ε, καταστραφεί ε, πάνω από 50 κτίρια στην ε, Βιέννη. Και πραγματικά σιγά σιγά με, την, με το χτίσιμο νέων σύγχρονων κτηρίων καταστρέφεται ο γνωστός παραδοσιακός χαρακτήρας της Βιέννης και οι πολίτες της αυτό δεν το θέλουν. Ευχαριστώ. Um, σε σχέση με τα που κύριος Μόντες ε, ένα σχόλιο για το θέμα της τοπικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης πέθρου. Πολλές από τις ε, δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία της πολιτικής κληρονομιάς ή της ε, φυσικής κληρονομιάς έχουν ως στόχο αυτό ακριβώς. Το πρόγραμμα αυτό των διαδρομών έχει το συγκεκριμένο στόχο δημιουργία συγκεκριμένων διαδρομών σε τοποθεσίες που είναι λίγο γνωστές έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εργαστούμε επί τόπου και να αναπτύξουμε αυτή την τεχνογνωσία αυτό το απαραίτητο know-how για να προβάλλουμε όχι μόνο την ίδια τοποθεσία αλλά και την γύρω περιοχή. Για παράδειγμα στην Αραγχουέθ στην Ισπανία. Η Αραγχουέθ και η περιοχή της Λαγκράνχα δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτά τα δύο, αλλά είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Είναι στην ίδια ζωτική περιοχή. Αυτές οι συνέργειες λοιπόν μπορούν να δημιουργηθούν μέσω αυτών των προγραμμάτων σε πολλά επίπεδα. Πολιστική βιομηχανία, πολιτική κληρονομιά, τουρισμός κλπ. κλπ. Έτσι ώστε να δοθεί μια όθηση, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή την πολιτική κληρονομιά για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της γύρω περιοχής. Η καινούρια έκθεση ανάπτυξης ε, του αστικού πολιτιστικού μέλλοντος αναφέρεται σε αυτό ακριβώς. Μιλάμε για μέλλον σε πόλεις γιατί ε, στο μέλλον σχεδόν όλοι μας τα ζούμε σε πόλεις. Αλλά ε, το, αυτή τη στιγμή γίνονται πολλές συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Κομισιόν για το πώς μπορούν να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών μέσω της πολιτικής κληρονομιάς. Νομίζω ότι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, για παράδειγμα, εστιάζεται, εστιάζει και σε αυτό. Οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω της δημιουργίας και της προστασίας προς της πολιτικής κληρονομιάς. Και μετά ήθελα να μιλήσω σε σχέση με τα όσα είπε ο, ο νομικός ο, ο, ο, νομικός συνάδελφος και εγώ είμαι νομικός το πλαίσιο των στόχων της χιλιετίας ε, μας αφορά όλους και όταν λέω όλους εννοώ όλους από τον πιο μικρό καθημερινό πολίτη μέχρι το, το τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς επίσης και το διεθνές UNESCO κλπ. κλπ. Ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Γιατί εμείς έχουμε αρμοδιότητα στην εφαρμογή των στόχων της χιλιετίας και μιλούμε για παράδειγμα για τον 11 και στο σημείο 4 λέει ότι θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να προστατέψουμε το φυσικό και πολιτιστικό ε, περιβάλλον. Ε, συγγνώμη, την ε, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του κόσμου. Του κόσμου. Και ε, αυτό είναι δουλειά όλων. Η δική σου, η δική μου, των παιδιών μας, όλων. Οπότε η προστασία της πολιτικής ισονομιάς έχει σχέση με τον καθέναν από εμά, με την καθεμία από, μια, Θα πρέπει να φύγουμε, να βγούμε από το κοινοβούλιο και να πάμε στους νέους, στους millennials, στου youtubers. Θα πρέπει να τους μιλήσουμε στην καρδιά τους με την πολιτική χρονομία γιατί αλλιώς το χάσαμε το παιχνίδι. Αλλιώς η πολιτική μας κληρονομιά δεν θα φτάσει στην επόμενη γενιά, θα μείνει σε εμά. Και αυτό πραγματικά είναι ομό που λέω, το έχω ξαναπεί, αλλά αυτή τη χρονιά, το 2018, πρέπει να κινήσουμε όροι. Γιατί ε, έχουμε μια κινητοποίηση εξαιτία χάρη σε αυτό το, χρόνο, το έτος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας χωρίς ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η κουλτούρα, ο πολιτισμός είναι κατακαιρματισμένος. Θα πρέπει όμως όλοι μαζί να συσπηρωθούμε. Ε, οι τοπικές αρχές, οι ευρωπαϊκές αρχές, οι περιφερειακές αρχές, όλοι. Και ο Διακόνου σίγουρα κάποιες από αυτές τις ιδέες τις συμμερίζεται. Ε, ε, είμαστε και οι δύο εξίσου παθιασμένοι. Αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω. Είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά θα πρέπει να βρεθούμε σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Εγώ ε, πρέπει να πω ότι τοποθετήκατε πολιτικά θα έχουμε και σύντομα τις εκλογές. Καλή σα ε, επιτυχία. Ζητώ συγγνώμη ε, να μην μιλάμε όλοι μαζί, λέει ο Πρόεδρος. Κλάου Πέτερ Έχτερ, μέλος ε, της Europa και το προηγούμενο μέλος που μίλησε, και αντιπρόεδρος της Europa από τη Γερμανία. Ως αντίκτυπος της πολιτικής κληρονομιάς υπόθηκε ε, νομίζω ότι τα όσα ακούστηκαν είναι πραγματικά σημαντικά, ε, σημαντικές επιτυχίες γιατί αύξησαν την ευαισθητοποίηση για την ε, πολιτική κληρονομιά και ε, επικεντρωθήκαμε κυρίως στο θέμα της βιωσιμότητας. Αλλά θα πρέπει να γίνουν κι άλλα, να γίνουν πολλά περισσότερα. Αν θυμάμαι, έγινε ένα φόρουμ, πολιτικό φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και συζητήθηκαν οι ε, στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης ε, και το 11.4 περιλαμβάνει την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά αυτό δεν ε, συζητήθηκε ενδελεχώς γιατί δεν κατάλαβαν προφανώς η πολιτική τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το μέλλον της πολιτιστικής κληρονομιάς Και αναφέρθηκε και το σχέδιο ε, δράσης, το να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική, την ορμή. Θα μπορούσατε να προσθέσετε κάποιες πληροφορίες παραπάνω για αυτό το ε, σχέδιο δράσης, για να το ξέρουμε κυρίως για το μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, Έρχομαι από το Κυπριακό Κοινοβούλιο και θα ήθελα για λίγο να αναφερθώ ή να δώσω, μια συνέχεια στο ερώτημα προηγουμένως που έχει τεθεί ποιος φέρει την ευθύνη όχι μόνο στις περιοχές όπου υπάρχει κράτος δικαίου και λειτουργά σωστά ένα σύνταγμα αλλά κυρίως στις περιοχές των κρίσεων. Εκεί δημιουργείται ένα πρόσθετο πρόβλημα όπου κανείς δεν είναι υπεύθυνο για τίποτα. Στη δική μου την πατρίδα, στην Κύπρο, ε, βιώνουμε μια κατάσταση όπου η πολιτιστική κληρονομιά, κινητήρια, εκκλησίες ή και άλλες αρχαιότητες ακόμα περνούν μέσα από μια ταλαιπωρία, δεν ε, τους έχει τύχει κανένας σεβασμός από τις κατοχικές αρχές. Αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σύντομο χρονικό διάστημα σε ένα πλήρη αφανισμό στην Κύπρο σε λίγα χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχουν τα μνημεία εκείνα τα οποία είτε ο χρόνος θα τα ξεπεράσει είτε η κακοδιαχείριση είτε από ανθρώπους είτε από παράνομες αρχές. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή της σε ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης ή διάσωσης κάποιων μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων, 25 στο σύνολο, και εδώ είναι και η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπλακεί πέραν των πολιτικών που έχουν αναφερθεί προηγουμένως ακόμα και στον τομέα της ανάληψης πρωτοβουλειών για ειρήνευση σε κάποιες περιοχές. Η εμπλοκή και η χρήση μέσων με σκοπό πάντοτε να χρησιμοποιήσουμε ή να διαμορφώσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ δύο πλευρών είναι πάντοτε ένα χρήσιμο εργαλείο. Και τον DG External ή η Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων θα πρέπει να είναι πάντοτε ιδιαίτερα προσεκτική εκεί και όπου δίνεται οικονομική βοήθεια αυτή η οικονομική βοήθεια, η διαχείρισή της θα πρέπει να της γίνεται με τέτοιον τρόπο που να μην θέτει σε κανέναν κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά. Δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται αναπτύξεις ή άλλα προγράμματα και η πολιτιστική κληρονομιά να τίθεται σε κίνδυνο. Όμως θα το επαναλάβω ότι αυτό ως εργαλείο η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν είναι ούτε στρατιωτική δύναμη, είναι μια πολιτική ένωση, είναι ένας οικονομικός οργανισμός, μια οικονομική δύναμη. Έχει αυτή την ευχαίρεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να το πράξει. Στην περίπτωση της Κύπρου όλα αυτά τα μνημεία οι αρχαιολογικοί χώροι που περιμένουν προστασία και διάσωση, επαναλαμβάνω διάσωση, έχουμε την υπεύθυνο, τους υπεύθυνους ποιοι είναι, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ να αναλάβει διάφορα προγράμματα. Και πάνω απ' όλα ποιο είναι ο υπεύθυνο, ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί σε αυτές τις περιοχές που πρέπει να αναπτυχθούν πάνω σε μόνιμη βάση, προκειμένου να υπάρχει επιτήρηση και επίβλεψη, είναι και ο ρόλος της UNESCO, είναι όμως και ο ρόλος και του Ευρωκοινοβουλίου με ψηφίσματα πάμπολα τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να υλοποιηθούν. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να, να πω ότι ο χρόνος σε αυτές τις περιοχές δεν είναι πάντοτε ο σύμμαχός μας και επανέρχομαι στο αρχικό θέμα της αναγκαιότητας για ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από την ψηφιοποίηση μπορούμε να καταγράψουμε κάτω αυτά τα μνημεία και τουλάχιστον να τα σώσουμε στους αιώνες των αιώνων. Ναι, οι δομές της οργάνωσης είναι πολύ σημαντικές που μπορούμε να αναλάβουμε και πολύ συχνά αυτές οι αρμοδιότητες είναι εθνικές αρμοδιότητες, όπως είπατε και εσείς. Παρακαλώ, κυρία μου, εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε για δεύτερη φορά ε, το λόγο. Νομίζω ότι όλα αυτά που λέμε εδώ θα έχουν αντίκτυπο στο μέλλον αν μπορέσουμε να επιλύσουμε δύο προβλήματα. Πρώτον, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση. Αν δεν μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τις επόμενες γέννες για τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Ένας ε, συνάδελφος νωρίτερα είπε ε, για τις προτιμήσεις που διαβιβάζουν οι γονείς στα παιδιά τους σχετικά με την επαγγελματική τους ειδίκευση. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης, θα πρέπει να μπορέσουμε να, να τοποθετήσουμε, αν θέλετε, τη διάσταση της πολιτικής κληρονομιάς στις πολιτικές τοποθετήσεις. Καμία από τις τοποθετήσεις που ακούμε δεξιά και αριστερά σήμερα στα κοινοβούλια και αλλού δεν αναφέρονται στο θέμα αυτό δεν φαίνεται να είναι υψηλής προτεραιότητας θέμα για τους πολιτικούς ηγέτε. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να το τοποθετήσουμε στα μηνύματά μας, τα πολιτικά. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσουμε για την διοργάνωση της συνάντησης αυτής και την πρόσκληση ενδιαφερομένων φορέων όπως και εγώ και τη δυνατότητα συζήτησης με εκπροσώπους των κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό να συζητούμε μαζί τους γιατί είναι θέματα εθνικής αρμοδιότητας. Εγώ εκπροσωπώ ενώσεις ενώσεις ειδικών που ασχολούνται με την ιστορική κληρονομιά, αν καταλαβαίνουμε καλά την ομιλήτρια, είναι πολύ σημαντικό γιατί μεγάλο ποσοστό των συνολικών μνημείων βρίσκονται σε ε, χέρια ιδιωτικών φορέων αρμοδίων που τα διαχειρίζονται και όταν μιλούμε για θέματα αποκατάστασης και συντήρησης κτηρίων είναι και αυτό μια καθημερινή ανησυχία και πολύ συχνά λείπουν, λείπει και η χρηματοδότηση, η οικονομική στήριξη της προσπάθειας αυτός. Νομίζω ότι μέσω της ε, φορολογικής πολιτικής θα μπορούσε να βρει κανείς ε, έναν τρόπο υποστήριξης τη της προσπάθειας της αποκατάστασης και συντήρησης των κτηρίων αυτών. Υπάρχουν πολλά εργαλεία που είναι στην εθνική εργαλειοθήκη, που είναι θέματα εθνικής αρμοδιότητας, προκειμένου να βοηθηθούμε να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, μπορώ να σας πείσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παθιασμένοι άνθρωποι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα που θα τους δοθούν. Οι εκπρόσωποι από την Ισπανία αναφέρθηκαν στην Ήπεθρο που είναι πραγματικά ένα θέμα κλειδί Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους τοπικούς υπευθύνου. και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσω πολύ συχνά απλών εργαλειών, απλών μέσων, αλλά χρειάζεται μια στήριξη, μια οργάνωση, δηλαδή απευθύνω μια έκκληση προς όλους τους υπευθύνους των κρατών μελών να τα προσέξουν αυτά τα στοιχεία. Και τέλος, συζητήσαμε για νομικό πλαίσιο και νομική βάση. Είναι σημαντικό αυτό γιατί και εγώ δικηγόρος είμαι αλλά υπάρχουν πάρα πολλά νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αντίκτυπο επί των μνημείων των πολιστικών και τα της ενεργειακής απόδοσης για παράδειγμα διότι έχουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις στους ιδιοκτήτες των κτηριακών συγκροτημάτων Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν στα νομοθετήματα τα ευρωπαϊκά που έχουν αντίκτυπο επί των πραγμάτων αυτών. Ε, βεβαίως πάντοτε υπάρχει αμφισημία και υπάρχει δυσκολία να εξασφαλίσουμε μια σωστή προσπάθεια. Και να ευχαριστήσω και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξετάζει τα θέματα των ιδιωτικών διαχειριστών εμείς μέσω μιας πρόσφατης μελέτης ε, εξετάζουμε business models σχετικά με την καλύτερη, την χρηστή διαχείριση γιατί όπως είπατε και εσείς κρύβονται άνθρωποι πίσω από όλα αυτά τα προγράμματα και τις προσεγγίσεις. Παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Um, Ευχαριστώ πολύ. Η δική μου παρέμβαση θα είναι πολύ σύντομη γιατί η συνάδελφος είπε τα περισσότερα που ήθελα να πω. Άννα Ρωμανόφσκι από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συντηρητών, Οργανώσεων Συντηρητών. Έχουμε μέλη σε 22 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη Να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν για την αναλογία που μας έκανε τη σύγκριση με τους γιατρούς γιατί είναι πολύ δύσκολο να ε, περιγράψει κανείς τι κάνει ένα συντηρητής. Είναι πολύ ιδιαίτερο ε, επάγγελμα. Να προσπαθήσω εγώ να εξηγήσω λίγο περί τίνος πρόκειται. Μιλούμε για αποκατάσταση και συντήρηση και πέραν της τέχνης παίρνει κανείς το καλλιτεχνικό, την καλλιτεχνική παραγωγή ενός αντικειμένου, παίρνει την καρδιά του ουσιαστικά. Αλλά το θέμα είναι να πουλήσει αυτό το, να προωθήσει αυτό το προϊόν. Και εκεί παρεμβαίνει ο συντηρητής για να το βελτιώσει, για να μπορέσει να προωθήσει το προϊόν αυτό. Και επειδή ακριβώς μιλούμε για τις παρεμβάσεις, τις άμεσες παρεμβάσεις, Υπάρχουν πολλές οριζόντιες προσεγγίσεις, ας πούμε για την πρόσβαση, γιατί χρειαζόμαστε τις κοινότητες. Πρέπει να γνωρίζουν οι κοινότητες την αξία της δουλειάς που κάνουμε. Αντιμετωπίζουμε πολλά εμπόδια όταν δουλεύουμε και δεν υπάρχει λύση. Οπότε το θέμα είναι θέμα έρευνας. Εμείς στην καθημερινή μας δουλειά αντιμετωπίζουμε πολλά τέτοια προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν η ευκαιρία, μια που είναι εδώ οι εθνικοί εκπρόσωποι, να το συνειδητοποιήσουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία για την, μέσω της αποκατάστασης και της συντήρησης των έργων τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορεί να βοηθήσει και στη βιωσιμότητα και στην επαναχρησιμοποίηση των ιστορικών μνημείων. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σημαντικούς εταίρους για την πολιτιστική κληρονομιά. Κάποιος είπε πιο πριν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τα εργαλεία για να παρέμβει. Εσείς οι εκπρόσωποι των κρατών μελών επίσης έχετε πολλά ε, εργαλεία στα χέρια σας με τους εμπειρογνώμονες, με τους ε, εμπλεκόμενους φορείς, γιατί είναι ειδικοί και γνωρίζουν. Οι συντηρητές αναλαμβάνουν πραγματικά μεγάλη ευθύνη για την προστασία του υλικού και των μνημείων. Προσπαθούμε λοιπόν από, από κάτω προς τα πάνω να παρέμβουμε. Προσπαθούμε να, κάνουμε, να είμαστε η ενδιάμεση με την κοινωνία. Αλλά ακόμα και σήμερα οι κοινωνίες μιλούν για ανθρωπογενείς καταστροφές. Κυρίως όταν μιλούμε για την αποκατάσταση και τη συντήρηση, γιατί οι πολίτες δεν, γνωρίζουν. Και επίσης δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για την αποκατάσταση και τη συντήρηση. Και καμιά φορά μας παρεξηγούν, δεν θεωρούμαστε εταίρο σε τέτοιου είδους συζητήσεις για τη διατήρηση της πολιτικής κληρονομιάς. Οπότε έχετε το και αυτό υπόψη. Υπάρχει μεγάλη προστιθέμενη αξία από τη δική μας τη δουλειά και δείτε το από νομική πλευρά και τι μπορείτε να κάνετε για να μας θεωρήσετε και εμάς ως έναν από τους εμπλεκόμενους φορείς σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Σύντομη η παρέμβασή σας. Άλλος κανείς που να μην είδα, που να θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε, που μας δίνετε το λόγο. Πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει την έδρα του στο Στρασβούργο, 47 μέλη και βασίζεται στις αρχές ε, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας. Εδώ και κάποια χρόνια εργαζόμαστε επί του θέματος του φυσικού και, της φυσικής και πολιτικής κληρονομιάς, ε, των τοπίων μέσω διεθνών συνθήκων που υπογράφονται, μονογράφονται, υπογράφονται από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και εφαρμόζονται από αυτά. Ε, όλο αυτό το κεκτημένο είναι πολύ σημαντικό να υιοθετηθεί από όλα τα κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης Ενδεχομένως μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να καταστεί συμβαλόμενο μέρος ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, υιοθέτησε την οδηγία για, ε, ε, για τα οικοσυστήματα με βάση την ε, σύμβαση της ε, Βιέννης ε, για την άγρια φύση, στην οποία έγινε συμβαλόμενο μέρος, της Βέρνης, συγγνώμη, για, το, για την άγρια φύση αλλά και της, ε, υπάρχει και η σύμβαση της Γκρενόμπλ για την αρχιτεκτονική κληρονομιά, της Βαλέτας για την αρχαιολογική κληρονομιά και η σύμβαση του Φάρο για τις αξίες ε, της ε, πολιτικής κληρονομιάς για την κοινωνία. Και σε αυτές θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει συμβαλόμενο μέρος. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία με την Κομισιόν, διοργανώνει επίσης Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτικής κληρονομιάς, με τεράστια επιτυχία ανοίγουν τις πόρτες τους μια σειρά από κτίρια, γίνονται επισκέψιμα για ένα χρονικό διάστημα και δεν μιλούμε μόνο για τα ενσώματα αγαθά αλλά και για άλλα αγαθά. Σε ό,τι διαφορά το, τη σύμβαση για το τοπίο, 39 κράτη ναι, έχουν υπογράψει. Έχει εμπνεύσει πολύ ενδιαφέρον γιατί αφορά όχι μόνο τα ιδιαίτερα τοπία, αλλά και τοπία που είναι πιο κοινά και μέσα σε πόλεις, αλλά και εκτός αστικού του. Η Επιτροπή Υπουργών προσφάτως υιοθέτησε μια σύσταση για τη συμβολή αυτής της διαδικασίας στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και στην βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Είμαι από την ε, Πολωνία, Πρόεδρε. Εδώ και 30 χρόνια συμμετέχω σε τέτοιου είδου συναντήσεις, συνεδριάσεις. Μιλάμε για την για τον πολιτισμό και το πώς επηρεάζει την Ευρώπη από πολύ πριν ενταχθεί η Πολωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούω λοιπόν όσα λέτε με πολύ χαρά, αλλά θα ήθελα από αυτήν την ημέρα να βγει κάτι απτό και να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για την συνεργασία μας. Θέλω να μιλήσουμε για πράγματα συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, μιλώντας για θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Προφανώς αυτό είναι αρμοδιότητα των πιο χαμηλών επιπέδων της ιεραρχίας, των τοπικών κοινοτήτων κλπ. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενδιαφέρει ένα βιβλιοθηκάριο, ένα διευθυντή μιας βιβλιοθήκης. Ε, η εκπαίδευση έχει σχέση με την εγκύτητα προς την τοπική κοινωνία και προς τους πολίτες. Η Πολωνία, χάρη στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες συντήρησης και διατήρησης των μνημείων της Πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που ωφελούνται και πώς. Για παράδειγμα, έχουμε κονδύλια για, την, ανακαινήσεις. Χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους κονδύλια, τέτοιου σηματοτήσεις. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η κατάσταση σε άλλες χώρες. Το, το επάγγελμα του συντηρητή Ποιο είναι το στάτους του σε άλλες χώρες. Είναι ένα καλό επάγγελμα. Η σημαία του, της Μαζέπα που έχει σχέση με την επανάσταση των Ουκρανών στο 17ο αιώνα ε, ε, επιδιορθώθηκε και συντηρήθηκε με τη βοήθεια Πολωνών συντηρητών. Ε, είναι σημαντικό να διευκολύνουμε τέτοιου είδους συνεργασίες. Εμείς έχουμε πολλές γνώσεις, ε, πολλή τεχνογνωσία και θα πρέπει να είναι δυνατόν να τη μοιραστούμε. Θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα μόνο αν συνεργαστούμε και μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές. Ευχαριστώ. Mai vrea cineva să intervină? Άλλος κανείς θέλει το λόγο? Παρακαλώ. Τελευταία παρέμβαση. Ζητώ συγγνώμη που επανέρχομαι, Πρόεδρε. Αλλά νομίζω ότι και ο κύριος Οριόλ και η εκπρόσωπος τώρα του Συμβουλίου της Ευρώπης το καθιστούν απαραίτητο. Συμφωνώ με τον κύριο Οριόλ. Υπάρχουν χώροι και είναι απαραίτητο και πολύτιμο να προστατευτούν. Αλλά προστατεύοντας παράλληλα ένα πολύ συγκεκριμένο στοιχείο πολιτιστικής κληρονομίας. Μπορεί να είναι ένα κάστρο, μπορεί να είναι ένα κτίριο άλλο, αλλά χρησιμοποιώντας και το προηγούμενο παράδειγμα της ιατρικής, πρέπει να κάνουμε μια διάγνωση. Η αποκατάσταση ενός συνολικού τοπίου είναι πιο περίπλοκο θέμα. Δεν είναι απλώς το θέμα της αποκατάστασης της ηλικής ενωστηρίου. Γιατί εκεί πρέπει να αποκαταστήσουμε έδαφος σε άλλο επίπεδο. Και η πιο σημαντική κληρονομιά είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν μπορούμε να δράσουμε αποτελεσματικά για την πολιστική κληρονομιά εάν δεν προστατεύσουμε τις πολύτιμες εκείνες δεξιότητες και την οικονομική δραστηριότητα των πολιτών που καλούνται να ζήσουν και να προστατεύσουν αυτά τα μνημεία. Μάλιστα, έχουμε έναν τελευταίο ε, παρεμβαίνοντα από την... Ε, ε, μάλλον τον κύριο... Ναι, Πρόεδρε, σχετικά με την αξιοποίηση της υπαίθρου μέσω του Natura 2000 και για την πολύ σημαντική ενεργειακή μετάβαση. Από την Charon Maritime που είναι μια πολύ σημαντική περιοχή που εντάσσεται στο Natura 2000 έχουμε καθημερινά ένα νέο έργο αιωλικών ή φωτοβολταϊκών πάρκων που πολύ συχνά ε, αντιμετωπίζουν πολύ ε, οργανωμένες έντονες αντιστάσεις ε, ενώσεων κατοίκων διότι προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον, το περιβάλλον του οικοσυστήματος, αλλά από την άλλη μεριά ε, αδειοδοτούμε έργα που έρχονται σε αντίθεση προς όλα αυτά. Και ίσως αν κάτι πρέπει να αναπτύξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σήμερα είναι να θέσουμε ένα πλαίσιο ευρύτερο σχετικά με, την ενεργειακή αυτή μετάβαση που, που είναι απαραίτητη για εμάς πλέον ιδιαίτερα για περιφέρειες ε, που έχουν μείνει λίγο πιο πίσω και σχετικά με έργα που πολύ συχνά διοδοτούνται σε συνθήκες, ε, πώς να πούμε, αντιφατικές. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα και στη Ρουμανία με ευρωπαϊκά κονδύλια. Μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε ε, κτίρια από το 14ο-15ο αιώνα. Δέκα μέτρα πιο κάτω υπήρχε άλλου είδους ευρωπαϊκή επένδυση. Ε, αλλά μιλούμε για ε, χωματερές και όλα κατάφεραμε να τα αναπτύξουμε, προσπαθώ τώρα να σας δείξω το φάσμα των επενδύσεων, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, λοιπόν, κάποια συμπεράσματα μετά την ε, συζήτηση. Η βοηθός μου έχει σημειώσει όλες τις ε, παρεμβάσεις, τις προτάσεις και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και τα συμπεράσματα για αύριο για την Ολομέλεια. Παραδέχομαι ότι θα ήθελα να είχαμε κάτι συγκεκριμένο, κάτι απτό μετά τη σημερινή συζήτηση. Ξέρετε ότι φέτος γιορτάζουμε το έτος της ε, πολιτιστικής λερομιάς και θα με ενδιαφέρε περισσότερο το feedback για αυτή τη χρονιά. Το δικό σας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίσατε, το τι θέλετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως σας ε, ευχαριστώ όλους τους ε, εμπειρογνώμονες και τους νομικούς για τις παρεμβάσεις, γιατί πραγματικά ε, μας βοήθησαν πολύ να καταλάβουμε πώς ε, διαχειρίζεται το κάθε κράτος μέλος ε, τον πολιτισμό. Και βεβαίως ε, είπαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει συστάσεις, προτάσεις, αλλά δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να ολοκληρώσει ή να ξεκινήσει κάποιο project. Οπότε εμένα θα με ενδιαφέρει να μου πείτε σε ποιο βαθμό αυτό, αυτή την ευκαιρία που σας δίνετε από το έτος πολιτιστικής κληρονομίας τη χρησιμοποιήσατε ως θετική ευκαιρία για τη χώρα σας και αν μπορέσει το έτος αυτό να αποτελέσει απάντηση σε κάποιο κάποια ερωτηματικά. Εμείς κάναμε κάποιες επισκέψεις σε διάφορα κρατημέλη και σε κάποια μέρη πραγματικά δόθηκαν πάρα πολύ καλές λύσεις σε προβλήματα, έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που χάρη στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής πολιτιστική κληρονομιά κατάφεραν να γίνουν πραγματικότητα. Ακούστηκαν πολύ σημαντικέ παρεμβάσει, πολύ σημαντικέ ιδέε υπάρχουν πραγματικά απτά προβλήματα που μας αναφέρατε και όλα θα τα λάβουμε υπόψη. Και ξέρω βεβαίως ότι έχετε απόλυτα δίκιο σε όσα είπατε. Εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια με τον πολιτισμό στην ε, Ρουμανία η δουλειά μου ήταν σχετική με τον πολιτισμό. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, πτυχές του πολιτισμού. Έχω ζήσει πολλούς δύσκολους καιρούς, πολιτικά, οικονομικά και μπορώ να δω τον πολιτισμό από διάφορες πτυχές. Είχα ζήσει τον πολιτισμό και κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περίοδου. Από το 90 και μετά καταλαβαίνω και την καπιταλιστική εκδοχή του πολιτισμού. αλλά και στο παρελθόν και τώρα πάντα αισθανόμουν ότι ο πολιτισμός είναι σαν ένα λουλούδι που βάζουμε στο πέτο η πολιτική. Το χρησιμοποιούμε για να δίνουμε καλή εντύπωση στους πολίτες. Αλλά όταν μιλούμε για χρήματα, όταν μιλάμε για κονδύλια, για προπολογισμό, ε, ο πολιτισμό πάντα παίρνει τα μικρότερα ποσά. Και αυτό δεν είναι σωστό. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικά συστήματα, πολιτικά, διοικητικά. Αυτό ισχύει για πολλά κράτη και κανείς δεν έχει καταλάβει ποτέ πόσο σημαντικό είναι ο πολιτισμό και η ιστορία συνολικά. Αν είσαστε Μάλλον εσείς ως μέλη της, ε, των Εθνικών κοινοβολίων θα μπορούσατε να αλλάξετε αυτή την οπτική, θα μπορούσατε να μεταφέρετε σωστά το μήνυμα για να υπάρξει ένας μοχλός πίεσης στα κράτη-μέλη, για να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η πολιτιστική κληρονομιά. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία στον πολιτισμό και στην κληρονομιά του. Ε, χρειάζεται να ενσωματωθεί ο πολιτισμός στην καθημερινότητά μας. Ο τομέας αυτός ε, συνδέεται με πολλά θέματα, με διάφορες πολιτικές, ε, με πολλές ε, γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες ασχολούνται. Είδατε πώς ε, παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλάμε για πολιτισμό. Υπάρχουν λοιπόν πολύ, συγκεκριμένοι δεσμοί σε διάφορους τομείς και αυτό πραγματικά είναι μια πολύ σύγχρονη προσέγγιση του πολιτισμού. Και αύριο βέβαια θα μιλήσουμε για τα θέματα αυτά, οπότε εσείς πρέπει να κάνετε τους αγγελιοφόρους των καλών προθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη. Το φθινόπωρο λέμε στην Ρουμανία ότι μετράμε τα κοτοπουλάκια που γέννησαν οι κότες για να δούμε πόσα είναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς τώρα, να μετρήσουμε τα αποτελέσματα των δράσεών μας. Και πρέπει βεβαίως και οι γραμμές του προϋπολογισμού να περιλαμβάνουν τον τομέα του πολιτισμού. Ε, πολλές φορές και στη βιομηχανία και στη γεωργία δίνονται πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι για τον πολιτισμό. Αλλά ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικό και εμεί προτείνουμε μια, μια σύγχρονη προσέγγιση. Και αύριο λοιπόν θα ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά και με τη νέα αυτή προσέγγιση. Ευχαριστώ όλους που με βοηθήσατε στη σημερινή συζήτηση. Δεν χρειάστηκε καν να χρησιμοποιήσω το σφυράκι μου. Οπότε μόλις μία φορά θα το χτυπήσω σήμερα, τώρα, για να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε λίγα λεπτά βεβαίως ακόμη και ε, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε και φωτογραφίες. Έχουμε 5-10 λεπτάκια, ε, μπορούμε να συνομιλήσουμε αν θέλετε, να σφίξουμε τα χέρια, μπορούμε να κλείσουμε την συνεδρίαση λοιπόν και τα λέμε αύριο.